Αξιότιμοι συνάδελφοι, ε, ξεκινάει και πάλι η συνεδρίασή μας. Μετά από το ε, μεσημεριανό φαγητό, ε, νομίζω είμαστε όλοι πιο... είμαστε ενωμένοι. Και τώρα έχουμε λοιπόν στο πρόγραμμα το επόμενο θέμα. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά εκείνον ο οποίος ε, είναι αρμόδιος ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους ε, στόχους μας αρμόδιος και για την συνεδρίαση Ρίο συν 20. Να εμφανιστούμε δηλαδή εκεί ενωμένοι ως Ευρωπαίοι και να παρουσιάσουμε μια καλή στρατηγική. Σας καλωσορίζουμε θερμά στην συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να έρθετε. Δεν θα ε, μακρηγορήσω άλλο. Θα δώσω ευθύς αμέσω το λόγο στον Επίτροπο και μετά θα κάνουμε αυτό που κάναμε και σήμερα το πρωί. Ε, ο κάθε μετέχων ε, θα έχει δύο λεπτά για την παρέμβασή του και θα κάνουμε πάλι το ίδιο. Δύο εθνικοί βουλευτές και μετά ένας ευρωβουλευτής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αξιότιμα οι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας μερικά πράγματα για την εξέλιξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας που μας οδηγεί στο Ρίο ΣΥΝ με χαροποιεί ιδιαίτερα που παρίσταμε εδώ σήμερα, γιατί πιστεύω ότι ο ρόλος, ε, το, ο κοινοβουλευτικός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο δικός σας ο ρόλος ε, μετά από το Ρίο θα είναι ακόμη σημαντικότερο Ελπίζουμε ότι οι κυβερνήσεις θα δεσμευτούν πλήρως ε, στο Ρίο τον Ιούνιο, αλλά τα κοινοβούλια είναι αυτά στα οποία λογοδοτούν οι κυβερνήσεις και πιστεύουμε ότι θα είστε καθοριστικοί στο να εξασφαλιστεί ότι οι δεσμεύσεις ε, μέχρι το Ρίο συν 40 δεν θα ξεχαστούν. Τρεις μήνες έχουμε ακόμη μέχρι τότε και πολλά πρέπει ακόμη να κάνουμε. Υπάρχουν ε, άτυπες συνεδριάσεις στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή ε, για την ε, προετοιμασία της διάσκεψης. Θα, θα γνωρίζετε ίσο ήδη την διαδικασία. Γνωρίζετε το πρώτο σχέδιο τελικού εγγράφου του Ιανουαρίου, ότι θα ληφθεί υπόψη οι συνεισφορές που ελήφθησαν, όπως επίσης και η δική μας συνεισφορά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γνωρίζετε ενδεχομένως τις αντιδράσεις που μερικές ήταν επικριτικές. Ήταν, είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις που θα έχουμε. Ήμουν την περασμένη εβδομάδα στο Ρίο Τζανέιρο και σε, μερικούς, σε μερικά λεπτά θα σας πω τη δική μου άποψη για την προετοιμασία ε, και την εξέλιξή της και τα ενδεχόμενα σενάρια. Πρώτον όμως θα ήθελα να εξηγήσω κυρίως για τους ε, ε, βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων πώς ε, εξελίχθηκε η δική μας ευρωπαϊκή θέση και πώς ε, η Επιτροπή διαμορφώνει την δική της προσέγγιση στην πράσινη οικονομία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρώπη η πράσινη οικονομία δεν είναι καινούρια ως έννοια. Όταν είχα την ακρόαση για να, ως υποψήφιος επίτροπος ανέφερα κάποια από τα στοιχεία της που θα πούμε ενδιέφεραν όλος ιδιαίτερος σε σχέση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, τότε δεν το είχα πει πράσινη οικονομία, το είχα πει ε, αποδοτικότητα των πόρων και τα τελευταία χρόνια αυτή αποτέλεσε ορόσημο της ε, ευρωπαϊκής μας στρατηγικής για το 2020. Αν ε, θέλετε να γνωρίζετε πώς βλέπει από την ευρωπαϊκή της πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πράσινη οικονομία, πρέπει να διαβάσετε το χάρτη πορεία για την αποτελεσματικότητα των πόρων, την αποδοτικότητα των πόρων που εγκρίναμε το Δεκέμβριο του 2011. Είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ευρύτερος στόχος ε, των πολιτικών είναι η αποσύνδεση της χρήσης των πόρων ε, και του αντίκτυπό και το αντίκτυπού της ε, στην ανάπτυξη. Αυτό χρειάζεται κάτι παραπάνω βέβαια από νομοθετική προσέγγιση. Χρειάζεται αλλαγές στη συμπεριφορά μας ως παραγωγών και ως καταναλωτών κάτι το οποίο με τη σειρά του σημαίνει ευρύτερη προσέγγιση πολλών, σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα οι περισσότερες από τις πολιτικές αυτές είναι στα χέρια εθνικών κυβερνήσεων και γι' αυτό η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου υπό ε, την Ευρώπη 2020 και ετήσια προγράμματα μεταρρύθμισης ε, είναι πολύ σημαντικό τμήμα. Θα ήθελα να ζητήσω από τους εθνικούς βουλευτές που παρίστανται εδώ ε, σήμερα να παρακολουθούν πολύ στενά τις ενέργειες των κυβερνήσεών τους σε σχέση με την ετήσια έκθεση ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2012 για παράδειγμα ζητήσαμε ε, τη μείωση των περιβαλλοντικών ε, ε, επιδοτήσεων και την μετάβαση στη σχετική φορολόγηση. Είναι ενδεχομένω μια ευρωπαϊκή προσέγγιση αυτή, όμως το πρόβλημα είναι ένα ε, παγκόσμιο πρόβλημα. Οι μεγάλες παγκόσμιες τάσεις καθιστούν ε, την ανάπτυξη πόρων ε, επιταγή. Είναι κάτι το αναπόφευκτο, είναι κάτι που πρέπει να γίνει και για τι χώρες που είναι πλούσιες και για τις χώρες που είναι φτωχές πόρους. Όλοι γνωρίζουμε ότι ε, θα είμαστε 9 δισεκατομμύρια στο μικρό μας πλανήτη μέχρι το 2005 και μέχρι τότε προβλέπεται ότι 3 δισεκατομμύρια επιπλέον ε, καταναλωτές ε, θα υπάρχουν. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τους 3 δισεκατομμύρια των οποίων το επίπεδο διαβίωσης θα αυξηθεί και για τις επιχειρήσεις βέβαια θα είναι σημαντικό γιατί θα ανθίσουν ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες τους όμως αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη πίεση στους πόρους και αυτή η πίεση θα είναι ο μεγαλύτερος περιοριστικός παράγοντας της ικανότητάς μας να αναπτυχθούμε ε, και να έχουμε ε, ε, υψηλό βιωτικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους πόρους, 140 δισεκατομμύρια περισσότερους, τόνους περισσότερους πόρους και είναι κάτι που θα παρουσιάσει αύξηση 70%. 60% του οικοσυστήματος μας, ε, ε, από το οποίο προκύπτουν οι πόροι αυτοί, υποβαθμίζεται. Μέχρι το 2030, αν δεν κάνουμε τίποτε, θα χρειαζόμαστε 40% νερό περισσότερο από αυτό ε, το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Ο αντίκτυπος της αύξησης κατανάλωσης θα είναι εκατοντάδες φορές μεγαλύτερος από την αρχή της εκβιομηχάνησης στην Ευρώπη. Ο πληθυσμός της Κίνας ε, σήμερα είναι 100 φορές ε, μεγαλύτερος ε, από αυτόν του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης. Και η Κίνα θα φτάσει σε επίπεδα ανάπτυξης σε μερικά χρόνια, τα οποία πήραν 100 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο να φτάσει. Μιλάμε λοιπόν για μια, ένα πραγματικό σοκ πόρων που θα είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερος και αυτό αφορά καθαρά την Κίνα και μόνο. Ε, η σπανιότητα πλέον των πόρων ε, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μεσαίας τάξης ε, θα περιορίσει την ανάπτυξή μας. Οι χώρες σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους πρέπει να προετοιμαστούν για την κατάσταση αυτή. Δυστυχώς το μήνυμα είναι το εξή και δεν είναι πολύ καλά κατανοητό μεταξύ όλων των διαπραγματευτικών μας εταίρων και κατά τον επόμενο μήνα η πρώτη μας πρόκληση θα είναι να εξηγήσουμε αυτήν τη λογική και να υπερβούμε την ε, υπόθεση ότι υπάρχει κάποιο ιδιωτελές ε, εγωιστικό κίνητρο πίσω από την πράσινη, πράσινη οικονομία, ε, όπως την αποκαλούμε. Έχω ακούσει πολλές θεωρίες συνωμοσία. ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ότι είναι μια προσπάθεια των πλούσιων χωρών ε, να περιορίσουν την ανάπτυξη των φτωχών χωρών ή να δημιουργήσουν ε, προστατευτικούς τείχους πράσινους ε, αυτή τη φορά. Πρόκειται για μια παρεξήγηση την οποία πρέπει να άρουμε γιατί ε, ο ανταγωνισμός έχει άμεση σχέση με τους ε, άλλους πυλώνες της αηφόρου ε, ανάπτυξης. Η πράσινη οικονομία είναι ένας από τους φορείς για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την αηφόρο ανάπτυξη και στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και όταν λέω αηφόρο ανάπτυξη εννοώ οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Θα εκτιμούσα όλο ιδιαίτερο την προσπάθειά σας για να περάσω αυτό το μήνυμα με κάθε ευκαιρία που θα έχω τον επόμενο μήνα ε, και ε, θα μπορούσατε να κάνετε και εσείς το ίδιο σε συναντήσεις με τους συναδέλφους σας. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής θέσης ε, για το Ρίο. Στις αρχές του μήνα, οι, αρχές, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Συμβούλιο ενέκριναν συμπεράσματα ότι πρέπει να κινηθούμε προς μένους επιχειρησιακού επιχειρησιακούς στόχους και ε, δράσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο Εντό συμπεφωνημένων χρονικών ορίων. Και αυτό ήταν μια παράθεση. Αυτό έδωσε πλήρη εντολή στου ε, υπουργού περιβάλλοντος ε, στο ε, Συμβούλιο για το Περιβάλλον πριν από 10, μήνες, 10 μέρες συγγνώμη, να δώσουν σάρκα και οστά σε ορισμένους τομεί που θα μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους αυτούς. Κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσει σε πέντε τομεί αρχή, του πυλώνες τη ζωή θα μπορούσαμε να του αποκαλέσουμε την αηφόρο ενέργεια, το νερό και ειδικότερα την αποδοτικότητα του νερού ε, υποβάθμιση της ε, γης ε, και, του, και των οικοσυστημάτων, ωκεανή και κάτι το οποίο είναι οριζόντιο είναι η αποδοτικότητα των πόρων και η επεξεργασία των αποβλήτων. Όλα αυτά πρέπει να ειδωθούν στο πλαίσιο της συνεισφοράς της πράσινης οικονομίας προς μια υφόρο ανάπτυξη και εξάλληψη της φτώχειας τα συμπεράγματα αυτά θα είναι ο βασικός μας ε, ε, γνώμονα στους ερχόμενους μήνες. Κινούμεθα ε, προ, προς την κατεύθυνση των πέντε αυτών τομέων που τόνισαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος. Βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ανησυχίες που αποτελούν προτεραιότητα άλλων διαπραγματευτικών εταίρων αλλά το επιχείρημα μας θα είναι ότι αν καλύψουμε αυτού τους πέντε πυλώνες θα καλύψουμε τις περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και τις ανάγκες μας από την αηφόρο πόλη μέχρι την αηφόρο γεωργία, από ε, την ε, ε, ασφάλεια των πόρων μέχρι την εξάλληψη της φτώχειας. Ε, οι ωκεανοί, το νερό, ε, η γη είναι πάρα πολύ απαραίτητα για την εξάλληψη της, πτω... της φτώχειας γιατί εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από οικοσυστήματα όπως ε, βοσκότοποι, όπως δάση για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Εν πάση περιπτώσει αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σε σχέση με την εξήγηση της αρχής αυτής ευχαρίστω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Κάτι ακόμη πρέπει να τονίσω. Το Ρίο Συν 20 είναι μια παγκόσμια διάσκεψη και δεν συμφωνούν βέβαια με, την, ε, με, τους, ε, με τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλοι οι εταίροι. Ε, αγωνιζόμαστε να φτάσουμε σε, στο φιλόδοξο αποτέλεσμα που πιστεύουμε ότι αξίζει στον κόσμο μας, όμως αυτό δεν είναι καθόλου εγγυημένο. Το πώς θα καταφέρουμε αυτό να συνάδει με την αρχή της αηφόρου ανάπτυξης ε, ε, και των σχετικών στόχων. Όπως γνωρίζετε, οι στόχοι, οι SDGs, οι στόχοι της αηφόρου ανάπτυξης είναι μια έννοια την οποία πρότεινε η Κολομβία και η Γουατεμάλα πριν από μερικούς μήνες ε, σε συνεργασία με την Βραζιλία που είναι πολύ σημαντικός εταίρος Τρία ε, σημεία θα ήθελα να θέξω για το πώς θα έπρεπε να αναπτυχθούν. Πρώτον, πρέπει να είναι ένα γενικό πλαίσιο για την κατάσταση μετά από το 2015 και την αηφόρο ανάπτυξη ε, με στόχους ε, που αντιμετωπίζουν βασικές προκλήσεις με πολύ σφαιρικό τρόπο. Να βασιστούμε δηλαδή στο, στην Ατζέντα 21, όπως επίσης και το πρόγραμμα δράσης, το σχέδιο δράσης του Johannesburg, ένα μείγμα μέτρων για να μπορέσουν μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, λύσεις που θα διαρκέσουν. Ε, δεύτερον, πρέπει να είναι πλήρω συμβατή με όλου του στόχου τη της πράσινη οικονομία. Και τρίτον, πρέπει να ε, είναι συντονισμένοι και να συνάδουν με του αναπτυξιακού στόχου τη χιλιετία και δεν πρέπει να ε, παρεκκλίνουν τι προσπάθειέ μα από την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων τη χιλιετία και την επίτευξη αυτών μέχρι το 2015. Αν υπάρχει λοιπόν μία διαφορά που είναι σαφή ανάμεσα στου στόχου τη αηφόρων ανάπτυξη και του αναπτυξιακού στόχου τη χιλιετία, αιτία είναι ακριβώς ότι οι δεύτεροι αφορούσαν κυρίω αναπτυσσόμενε χώρε, ενώ οι πρώτοι αφορούν κυρίω ε, δεσμεύσει για όλου, για όλε τι χώρε σε κάθε στάδιο ανάπτυξη και αν βρίσκονται. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία με τι υπόλοιπε χώρε, ε, ε, εμείς αξιολογούμε τις θέσεις των υπολείπων, ξεκινώντας με τη Βραζιλία ε, και την Λατινική Αμερική γενικότερα, να δούμε τι ε, κοινούς παρονομαστές μπορούμε να έχουμε για να υπάρξουν συμμαχίες και να, υπάρχει ένα, ε, να έχουμε ένα επιτυχές αποτέλεσμα στο Ρίο όλοι, όλες οι ανησυχίες όλων των υπήρων πρέπει να γίνουν κατανοητές και αν είναι δυνατόν ο στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να είναι να ε, ανοίξει ε, σταδιακά μια διαδικασία ε, πολυμερή διαπραγματεύσεων ώστε να υπάρξει σύγκληση και συνεργασία βάσει συγκεκριμένων θεμάτων και βάσει συγκεκριμένων περιφερειών και χωρών. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε το πλαίσιο του Ντέρμπαν ε, για να ε, επιτύχουμε μια ευρύτερη, πιο ανοιχτή διαδικασία. Ήδη γνωρίζουμε ότι κάποιες χώρε έχουν σοβαρές ανησυχίες για την πράσινη οικονομία. Οι ανησυχίες αυτές ε, επικεντρώνονται γύρω από τον πράσινο προστατευτισμό, νέους όρους, εμπόδια στο εμπόριο και προβλήματα για τα οικοσυστήματα και την βιοπικιλότητα. Όμω αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι το επίπεδο σύγκληση κατανόησης μεταξύ Αφρικανική Ένωση και της Ευρωπαϊκής Ένωση γύρω από το θέμα της πράσινης οικονομίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί οι περισσότερες πιο ευάλωτε χώρες ε, του κόσμου βρίσκονται σε αυτή την ε, περιφέρεια. Και όταν συζήτησα με τις χώρες αυτές, ε, στην Κένια, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης στο Ναϊρόμπι ότι αυτή είναι η στρατηγική τους επιβίωσης, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι το πραγματικά καλό. Υπήρξαν επίσης σοβαρές ανησυχίες για την κινητοποίηση επαρκών μέτρων ε, εφαρμογής για την διευκόλυνση της μετάβασης στην πράσινη οικονομία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί με ε, τους κατάλληλους τρόπους. Θα είναι ένα από τα σημεία που ε, θα επιζητήσουν ιδιαίτερη συνεργασία για σύγκληση σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο με την ομάδα G77, αλλά και με την Κίνα. Οι προκλήσεις αυτές ε, ζητούν ε, μεγαλύτερη προσπάθεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για συνεργασία και συντονισμό με τους εταίρους μας μέχρι την διάσκεψη του Ρίο. Είχα ήδη διμερείς επαφές ε, με ε, αρμόδιους υπουργού από τις διάφορες περιφέρειες ε, στην Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της διάσκεψης που έγινε το Φεβρουάριο. Επίσης πήγα στη Βραζιλία την περασμένη εβδομάδα όπως σα είπα και θα περάσουμε τώρα στη δεύτερη φάση επαφών για να προσπαθήσουμε να ε, λάβουμε υπόψη ε, τις ε, ανησυχίες βασικών χωρών. Παράλληλα θα δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ένας ενεργός ακροατής που έχει την ικανότητα να αντιδρά θετικά και να προσαρμόζεται, κάτι το οποίο είναι μια προϋπόθεση για να φτάσουμε στην επιτυχία από κοινού. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία τη συμμετοχή τη κοινωνίας των πολιτών ε, και των επιχειρήσεων μέχρι το Ρίο αλλά και μετά το Ρίο. Η συζήτηση που θα γίνει για την πράσινη οικονομία στο Ρίο συμπεριλαμβάνει ε, τον επιχειρηματικό τομέα ε, σε μεγάλο βαθμό και δίνει τη δυνατότητα θέσεων απασχόληση, ευημερία όπως επίση και μεταφοράς τεχνολογία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να συμφωνηθούν σαφείς στόχοι στο Ρίο. Θα δώσει ε, σαφή μηνύματα και στον ιδιωτικό τομέα για την μελλοντική αξιολόγηση των επιχειρήσεων, κάτι που θα βοηθήσει στην καθοδήγηση της παραγωγής προς την σωστή κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών θα ζητήσει μεγαλύτερη εφαρμογή της αρχής της ε, πρόσβασης πληροφορίες, ε, τη δημόσια ε, συμμετοχή, όπως επίσης και τη συμμετοχή του κοινού στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό να επιτύχουμε την την κοινωνική πτυχή, να μην μείνει η κοινωνική πτυχή εκτός της όλης προσπάθειας. Ακούσαμε επίση ότι ομάδες κοινωνίας των πολιτών και ενδεχομένως κοινοβούλια σε κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ανησυχίες και για την πράσινη ε, οικονομία. Και αυτό μπορεί να ισχύει για παράδειγμα για τη Βραζιλία και για τις ε, χώρες Λατινικής Αμερικής γενικότερα. Υπάρχει λοιπόν η ευκαιρία από, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια και ε, την ε, ΟΚΕ ή την Επιτροπή ε, των Περιφερειών να έρθουν σε επαφή με κάποιους από τους εταίρους τους και να συζητήσουν αμοιβαία συμφέροντα λόγω της πράσινης οικονομίας. Το γενικό μας μήνυμα πρέπει να είναι ότι η θέση μας για την πράσινη οικονομία λαμβάνει υπόψη ε, την κοινωνική ένταξη, λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικές πτυχές ε, και είναι μια ευκαιρία για όλες ε, τις χώρες σε κάθε επίπεδο ανάπτυξης. Έχουμε ένα θετικό πρόγραμμα να προτείνουμε. Η πράσινη οικονομία πρέπει να είναι ένα μέσο για να επιτύχουμε την αηφόρο ανάπτυξη. Ε, με όλες τις πτυχές, την οικονομική, την κοινωνική, την περιβαλλοντική, τους σχετικούς στόχους και μπορεί επίσης να δώσει ε, τη δυνατότητα εξάλληψης ε, της φτώχειας και έτσι επιστημιστικής ασφάλειας. Το Ρίο του 1992 ήταν ε, γεμάτο από φιλοδοξίες, ε, ε, ετοιμότητα να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο, ένα καλύτερο μέρος να ζει κανείς. Το 2012 δεν μπορούμε όμως να παραγνωρίσουμε τη σοβαρή οικονομική κρίση. Δεν θα μπορέσουμε επίσης να αδιαφορήσουμε για ορισμένα νέα στοιχεία βάσει της καλύτερης κατανόησης που έχουμε σήμερα πολλών προκλήσεων. Προκλήσεων που είναι κοινέ για όλους μας και που θα έπρεπε να μας συνενώνουν όλους στο Ρίο. Και αν υπάρχει λιγότερη, ε, λιγότερη αισιοδοξία ε, γύρω μας, ε, υπάρχει και θα υπάρξει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη να καταστήσουμε τον κόσμο έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννος Ποτόσνικ. Εδώ βρεθήκαμε για να συμβάλλουμε στην βελτίωση της ζωής ε, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν ζουν οι άνθρωποι. Έχουμε συναδέλφους εδώ από 20 κράτη-μέλη και ήδη έχω μια σειρά από συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο για τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, επαναλαμβάνω, <clears throat> παρακαλώ συμπληρώστε την κάρτα όπου ζητάτε το λόγο, θα έρθουμε να την πάρουμε από τη θέση σας. Για τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισχύει η συνήθιση διαδικασία, σηκώστε το χέρι. Και τώρα... Ο συνάδελφος Μπρίνκαρτ από την Μάλτα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ασχοληθώ με την πράσινη οικονομία. Αν θέλουμε να αποφύγουμε τις παγίδες και τα ταπεινώσεις των διαπραγματεύσεων για το κλίμα και αν θέλουμε απτά αποτελέσματα, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο για μια πράσινη οικονομία, αλλά και ένα χάρτη πορείας για μια πολυμερή και πολυπολική αλλά και εθνική προσέγγιση. Να διευκρινίσουμε Πώ θα ανταποκριθούμε στις τοπικέ ανάγκε πριν κάνουμε μαθήματα στους άλλους για το τι να κάνουν και πώ να τα κάνουν καλύτερα. Δεν είναι θέμα επιλογής μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ενό καθαρού πλανήτη. Και τα δύο πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. <clears throat> Ακόμη και ο ιδιωτικό τομέας έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. Αλλά δηλώσει προθέσεων δεν αρκούν. Θέλουμε πολιτικέ εφαρμόσιμες και οικονομικά εφαρμόσιμες επίσης. Αν θέλουμε να επιτύχει η πράσινη οικονομία, θέλουμε σωστούς δείκτες που να αξιολογούν σωστά και θέλουμε και στοιχεία που να μας επιτρέπουν να οριοθετούμε την πρόοδο που πρέπει να σημειώσουμε. Δεν υπάρχει μια συνταγή για όλα, δεν υπάρχει ένα μέτρο πανάκια. Γιατί πρέπει η πράσινη ανάπτυξη να είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της κάθε χώρας. Αλλά υπάρχουν και μερικές γενικές ανάγκες επί των οποίων πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε αντίθετα από τις διαφορές μεταξύ χωρών και περιφερειών. Πιστεύω λοιπόν πρέπει να απλοποιήσουμε και να εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη τα κύρια θέματα που απασχολούν την λεγόμενη στρογγυλή τράπεζα για την κλιματική αλλαγή. Αλλιώς δεν θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και κάτι τελευταίο. Χωρίς καλή διακυβέρνηση, η αηφόρος ανάπτυξη στα πλαίσια ιδίω μιας πράσινης οικονομίας δεν μπορεί να επιτύχει σε κανένα επίπεδο, διεθνές, τοπικό ή επιχειρηματικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκούντερ από τη Ρουμανία και είναι εκπρόσωπος του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να αδράξω την ευκαιρία για να χαιρετήσω τους συναδέλφους μου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στον αγώνα κατά της οικονομικής κρίσης. Για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης πριν από τη διάσκεψη του Ρίο. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Το είπαμε ήδη. Η Ρουμανία έχει αρκετά λυπηρή πείρα από τα αποτελέσματα διαπραγματεύσεων ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ξέρετε η Ρουμανία είναι πολύ ανοιχτή χώρα προς οτιδήποτε ευρωπαϊκό, προς τη συνεργασία γενικά. Ακόμη και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει προστασία της οικονομίας της. Και ωστόσο, ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώμα επέλεξε να μπλοκάρει την ένταξη της Ρουμανίας στο χώρο Σέγγεν. Γι' αυτό είμαστε αρκετά απεσιόδοξοι όσον αφορά αυτή τη διαδικασία διαπραγμάτευση, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Η μηδενική εκδοχή του κειμένου μπορεί να βελτιωθεί αν λάβουμε επίσης υπόψη την πείρα της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την ε, αηφόρο ανάπτυξη και του προγράμματο των ΗΠΑ για το περιβάλλον. Η επιτυχία τη 19 η Συνόδου τη Επιτροπής του ΟΗΕ που έγινε το Μάιο του 2011 για, υπό την Προεδρία της Ρουμανίας είχε επιπτώσει σε όλη τη διεθνή κοινότητα. Ήταν σημαντική συμβολή για την ε, προπαρασκευή του Ρίο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα προγράμματα που θα επιτρέψουν τη δημιουργία μας πράσινης οικονομίας. Ωστόσο, το τελικό έγγραφο από τη συνδιάσκεψη αυτή δεν συμπεριέλαβε μια τροπολογία που αφορά το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών, ιδίω των λαών που ζουν υπό ξένη κυριαρχία, όσον αφορά τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε μόνο εάν στόχος μας είναι μια πράσινη οικονομία που να συνδυάζεται με την καταπολέμηση της φτώχειας μέσω ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου. Πρέπει οι στόχοι να έχουν σφαιρικό χαρακτήρα, πρέπει να είναι εύκολα δημοσιεύσιμοι και να μην θίγουν την, τους στόχους της χιλιετίας. Όσον αφορά την συνάντηση κορυφής του Ρίο, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να αποτελέσουν τμήμα του πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης μετά το 2015. Να συνδυάζονται δηλαδή με τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης της χιλιετίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ακόμη κάτι άλλο. Η Ρουμανία θα επιμείνει σε δύο προτάσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στο κείμενο. Είναι προτάσεις που υποστηρίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντός μας. Πρόκειται για μια μόνιμη προσπάθεια πολιτιστικής ανάπτυξης της υπαίθρου, να, δημιουργήσουμε, να δημιουργήσουμε δηλαδή βιώσιμες ε, κοινότητες στην Ήπεθρο, σεβόμενοι τις εθνικές ιδιομορφίες των κρατών. Και δεύτερον, αναγνώριση της σημασίας της ειδικευμένης τεχνολογίας που επιτρέπει με βάση τις γεωδιαστημικές πληροφορίες που έχουμε στους λαμβάνοντες αποφάσεις να εφαρμόζουν όλες τις ενέργειες που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία των ε, φυσικών πόρων, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες ανάπτυξης των περιφερειών και των χωρών του κόσμου. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Γκέρμεν και Μπράντι τώρα. Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ρίο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όλοι ξέρουμε την ε, εταιρεία αυτοκινήτων BMW. Για όσους δεν ξέρουν, δύο από τα τρία αυτοκίνητα που προσπαθούν να σας προσπεράσουν ε, αναβοσβήνοντας φώτα όταν είστε στην αριστερή λωρίδα είναι BMW, είναι ισχυρά αυτοκίνητα και τα αγοράζει ο κόσμος γιατί τους αρέσει η επιτάχυνση και να κάνουν φιγούρα. Αλλά αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον. Κοιτάξτε τις διαφημίσεις της BMW. Δεν μιλάνε για ταχύτητα, επιτάχυνση ή για τις διαστάσεις ε, του αυτοκινήτου μιλάνε για τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακος και την κατανάλωση καυσίμων. Πολύ καλό παράδειγμα πώς η βιομηχανική επανάσταση που ζούμε αυτή τη στιγμή επηρεάζει τα πάντα. Η πράσινη ανάπτυξη, η πράσινη οικονομία δεν είναι κάτι που το αναπτύσσουμε εμείς εδώ ως πολιτική. Συμβαίνει ενώ μιλάμε. Οι επιχειρήσεις του αύριο ή θα είναι βιώσιμες ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή είναι κατά την άποψή μου η οικονομική πραγματικότητα. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό εμείς οι Ευρωπαίοι για να γίνουμε πολύ πιο ανταγωνιστικοί να έχουμε έναν πιο βιώσιμο, πολύ πιο βιώσιμο τρόπο ανάπτυξης. Αλλά σφαιρικά σημαίνει ότι πρέπει να πείσουμε και τον κόσμο και να προετοιμάσουμε τον κόσμο για κάτι τέτοιο. Ο Επίτροπος Ποτότσινη μίλησε για την έκρηξη των τιμών των πρώτων υλών. Μα αυτό είναι ένα από του κύριου λόγου που πρέπει να περάσουμε στην πράσινη οικονομία. Και αυτή είναι μία από τι προκλήσει του Ρίο. Να πείσουμε τι αναπτυσσόμενε χώρε ότι η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι κάτι που προσπαθούμε να επιβάλλουμε ω δυτικό κόσμο. Είναι κάτι που θα διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο και το δικό του μέλλον. Που θα είναι η πιο επιτυχή ανάπτυξη που θα μπορέσουν να σημειώσουν. Τώρα για την κατάληξη του Ρίο αν επιτύχουμε να πείσουμε γι' αυτό ακριβώς τι αναπτυσσόμενε τις αναπτυσσόμενες χώρες, αυτή η προσπάθεια πειθούς μπορεί να είναι σημαντικότερη από τα γραπτά πορίσματα. Αυτό είναι για μένα το στοιχείο κλειδί για την πράσινη οικονομία στο Ρίο. Σήμερα το πρωί, μετά την συνάντησή μας, είχα μια πολύ θετική εντύπωση. Πιστεύω ότι ως Ευρωβουλευτές και βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων έχουμε τις καλύτερες προθέσεις, αλλά δεν θα πρέπει απλώς να φύγουμε από αυτή τη συνεδρίαση και να μην αξιοποιήσουμε την ισχύ που έχουμε ως νομοθέτες. Και έχουμε το δίκτυο κοινοβουλευτικών Globe, θα συναντηθεί στο Ρίο το πρώτο Σαββατοκυριακό και θα ήθελα να πιστείτε κι εσείς ότι πρέπει να γίνετε μέλη αυτού του παγκόσμιου δικτύου νομοθετών και να το αξιοποιήσετε. Μπορούμε να ασκήσουμε έτσι περισσότερη πίεση στις κυβερνήσεις μας για να έχουμε καλύτερη κατάληξη του ρίου. Όπως ακριβώς και θέλουμε και ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Κέρβεν Γκεμπράντι, ένας παλιός γνωστός τώρα, ο συνάδελφος Αδάμου, που ήταν ευρωβουλευτής της ΓΚΟΕ και συντονιστή. Παρακαλώ, δύο λεπτά. Και πάλι ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την ε, εισαγωγή του ομιλία που κατάληξε στο να είναι αισιόδοξη. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο προηγουμένω στο Προεδρείο σας ο οποίος έφερε το παράδειγμα της BMW και φυσικά αυτό το πράγμα για την BMW ήταν μόνοδρομο, δεδομένου ότι για να πουλά αυτοκίνητα πρέπει να έχεις και πλανήτη. Άμα δεν έχεις πλανήτη, ούτε αυτοκίνητα θα πουλάς, ούτε τίποτα. Γι' αυτό και λογική η στροφή που έκαναν στο να διαφημίζουν για τις εκπομπές διεξιδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα τους. Αλλά η οικονομική κρίση, κύριε Πρόεδρε, που ταρανίζει τον παγκόσμιο και που έχει φέρει εκατομμύρια συνανθρώπου μα στα όρια τη οικονομική εξαθλίωση, καθιστά την ανάγκη επίτευξη αεφόρου ανάπτυξη ακόμα πιο επιτακτική. Δυστυχώ η παγκόσμια οικονομική κρίση, εκτό από τι οικονομικέ και κοινωνικέ τη επιπτώσει, πλήττει παράλληλα και τι προσπάθειε προστασία του περιβάλλοντο, αφού έχει οδηγήσει σε πολλέ περιπτώσει στην αποδυνάμωση των πιο φιλόδοξων προτάσεων για την προστασία του περιβάλλοντο και την αφιέρωση των πόρων που θα διετίθεντο για αυτέ σε άλλου τομεί. Είναι για τους λόγους αυτούς που κατά τη δική μου άποψη θα πρέπει να αναλυφθεί σοβαρή πρωτοβουλία στο διεθνές επίπεδο για την άμεση προώθηση της επίτευξης της πράσινης οικονομίας και της αϊφόρων ανάπτυξης στην επερχόμενη διάσκεψη του Ρίο. Η επίτευξη των στόχων της πράσινης οικονομίας, της αηφόρου ανάπτυξης και της εξάλληψης της φτώχειας απαιτεί πρωτίστως συντονισμένη αλλά ταυτόχρονα και αποφασιστική δράση στο διεθνές επίπεδο με καθαρούς στόχους και χρονοδιαγράμματα επίτευξης τους. Συνεπώς, για να καταστεί δυνατή υπεραιτέρω πρόοδο πρόοδος τους εν λόγω τομής, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ερχόμενη διάσκεψη του Ρίο θα πρέπει να πιέσει προς την κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας για την κατάκτηση, κατάκτηση ενός οδικού χάρτη για την πράσινη οικοδομία με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις στο διεθνές επίπεδο. Οι στόχοι για την αηφόρο ανάπτυξη που θα συμφωνηθούν θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και σε πλήρη συνέργεια τόσο με τους στόχους της χιλιετίας αλλά και με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη της αηφορίας. Κατά την άποψή μου, οι στόχοι για την ανηφόρο ανάπτυξη που θα καθοριστούν θα πρέπει να έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα και όπου είναι δυνατό να έχουν κοινέ διαδικασίες με τους στόχους της χιλιετίας που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει καθιονδήποτε καθιονδήποτε τρόπο να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης των εν λόγω στόχων. Τα μέτρα που θα υιοθετηθούν στο διεθνέ επίπεδο θα πρέπει επίση να έχουν σαν κύριου άξονε του την κοινωνική, πολιτισμική και την ανθρώπινη διάσταση τη ανάπτυξη, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλο τη κοινωνία των πολιτών και να ενδυναμωθεί η αποτελεσματικότητα τόσο των πολιτικών όσο και των μέτρων για να εξασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη και να καταπολεμηθεί η φτώχεια και η πείνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ιδάλγο τώρα. Από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω ότι συμμεριζόμαστε τις περισσότερες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ομάδας υψηλού επίπεδου των ε, Ηνωμένων Εθνών. Το πρωί είπα ότι η οικονομική κρίση είναι βέβαια κίνδυνος, αλλά είναι επίσης και ευκαιρία. Τώρα μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές που θα μας οθήσουν προς, προς ένα βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης. Ξέρουμε βέβαια το κόστος που έχει ένα μη βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την Ισπανία και τη διεκδικούμε. Οι πράσινες πολιτικές όπως η ανακύκλωση είναι επίσης δυνατότητα δημιουργίας απασχόλησης και πλούτου. Βεβαίως πρέπει να μετατραπούν οι υποδομές όπως οι σιδηρόδρομοι για να ευνοηθεί η πράσινη οικονομία. Αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα. Πρώτον, η βιωσιμότητα έχει τιμή. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίσουμε ότι πρέπει να πουλήσουμε. Να το πληρώσουμε, συγγνώμη. Η ανακύκλωση, τα ανανεώσιμα, ο καθαρισμός των υδάτων, η διατήρηση των δασών, οικολογικά και υγιεινά τρόφιμα, η διατήρηση των οικοσυστημάτων στην Ήπεθρο και των ε, ατόμων έχει τιμή που πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να το πληρώσουμε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις μεταρρυθμίσεις, είτε της κοινή γεωργικής πολιτικής, είτε της αλληλευτικής πολιτικής, πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτά τα θέματα. Η κοινωνική βιωσιμότητα των πολιτικών. Και οι πολιτικές γεωργικών τιμών πρέπει επίσης να προσαρμοστούν γιατί πολλές φορές ε, την αυξημένη τιμή των καλύτερων προϊόντων ε, τις παίρνουν οι μεσάζοντες. Να διορθώσουμε λοιπόν τις ανισότητες, αλλά οι ανισότητες δεν είναι μόνο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν χώρες και περιοχές που χρειάζονται την αλληλεγγύη. Χρειάζονται μείωση των ανισοτήτων, γιατί έχουν χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. Αυτός πρέπει να είναι κοινό στόχος όλων των ε, συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Αντωνέσκου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκφράζω την ικανοποίησή μου που σήμερα συναντάμε τους ε, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια σε τελευταία ανάλυση είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την στήριξη και δημοσιοποίηση των μηνυμάτων αυτών στους πολίτες της Ευρώπης. Ήδη υπόθηκε συχνά ότι οι πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να είναι πολύ πιο αποφασιστικές, πρέπει να έχουν περισσότερο δυναμισμό, γιατί η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής είναι περιορισμένη. Πρέπει λοιπόν να δεσμευθούμε υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης. Και εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένους στόχους και τρόπους αξιολόγησης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίτευξης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο οικονομικός και ο κοινωνικός άξονας και όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος πρέπει να αποσυνδέσουμε την οικονομική ανάπτυξη από την υπερβολική χρήση πόρων και την βλάβη του περιβάλλοντος πράσινη οικονομία δεν μπορεί να επιτύχει παρά μόνο εάν συμμετάσχει και ο ιδιωτικό τομέα. Να ενθαρρύνουμε τι αγορέ και τι ιδιωτικέ επενδύσει, ούτω ώστε να συμμετάσχουν στην βιώσιμη ανάπτυξη. Και επίση να καταργηθούν όλε οι επιδοτήσει που μακροπρόθεσμα θίγουν το περιβάλλον. Και κάθε σημασία να δοθεί στη γεωργία. Και χρειαζόμαστε επίσης ένα κανονιστικό πλαίσιο σαφές, αξιόπιστο, που να δίνει στους οικονομικούς παράγοντες βεβαιότητα. Τα στοιχεία προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Και θέλουμε και συγκεκριμένους τρόπους χρηματοδότησης πιο ευφυείς. Να μην αγνοήσουμε, για παράδειγμα, τις εταιρικές σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όλοι όσοι δρούν στην οικονομία να έχουν νέα μέσα χρηματοδότηση διάθεσή τους και πιο συγκεκριμένα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάθε κανονιστικό όργανο θα επιτύχει εάν και μόνον εάν συνδυάζεται με εκστρατείες ενημέρωσης και εκστρατείες κατάρτισης. Μόνο έτσι πιστεύω ότι θα έχουμε ένα θετικό πολλαπλησιαστικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ η κυρία Βόλι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θέλω να μιλήσω λιγάκι για την πράσινη οικονομία και για το πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις σε, όλη αυτή τη διαδικασία. Και θέλω να κάνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δούμε κατά πόσον μπορείτε να οργανώσετε κάποιες εκδηλώσεις πριν από την συνδιάσκεψη κορυφής ε, το Ρίο. Οι επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη ίσως ε, μπορούν να ε, διευκρινίσουν λιγάκι την ατζέντα των πρώτων υλών, το τι έχει κάνει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε κατά πόσον η BMW και οι άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πόσο πράγματι κάνουν εξοικονόμηση γιατί αυτό δεν αφορά μόνο τον ανταγωνισμό αφορά και τον πλανήτη γενικότερα. Έτσι λοιπόν έχοντας αυτά κατά νου όπως επίσης και τα σχόλια των συναντέλφων, νομίζω ότι πρέπει να καλέσουμε όλα τα μέλη που βρίσκονται εδώ να προσχωρήσουν στο Globe ε, και θεωρώ ότι πριν από το Ρίο αυτό θα σημαίνει κάποια σημαντική διαφορά, γιατί θα είναι η ευκαιρία για τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετάσχουν στο λίγο για τελική ανάλυση. Εμείς καλούμεθα να νομοθετήσουμε και εκ των υστέρων να εφαρμόσουμε την νομοθεσία. Έχω επίσης μαζί μου πληροφορία για τις ε, κατακριμνήσεις. Ε, φαντάζομαι θα γνωρίζετε όλο το σχετικό τραγούδι και την έκθεση φωτογραφίας το τραγούδι το περίφημο του Bob Dylan για τη σκληρή βροχή, hard rain, να ξέρουμε τι ακριβώς έχουν οι άνθρωποι κατά νου. Να ληφθεί υπόψη στις πολιτικές διαπραγματεύσεις. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προάγει αυτό το project ε, μαζί με το Globe νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταστήσουμε σαφές τους ανθρώπους σε τι ακριβώς διακυβεύεται. Ότι είναι επίγον να αναλυφθεί δράση τώρα και ευθύ αμέσω μετά τη συνδιάσκεψη του Ρίου. Από την Ισπανία, ο συνάδελφος Απαρίτσου. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Δεν θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν το πρωί. Ισχύει νομίζω η πρόταση ψηφίσματος που μας υποβάλλατε. Θεωρώ ότι είναι καλή. Και για το θέμα που μας απασχολεί σήμερα το απόγευμα θέλω να επιμείνω σε δύο-τρία θέματα του ψηφίσματος αυτού που θέλουν πιστεύω περαιτέρω διευκρίνηση και επιμονή. Το βασικό λοιπόν είναι οι πόροι και τρεις τομείς ε, μας απασχολούν ενέργεια, είδωρ και απόβλητα. Βεβαίως είναι σημαντικό το είδωρ, αλλά όχι μόνο η ανάγκη χρήσης του, αλλά πολλές φορές και τα προβλήματα που υπάρχουν με την παροχή. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε να αποφύγουμε ε, την αλάτωση των ε, υδροφόρων οριζόντων γιατί δεν λαμβάνουμε αρκετή φροντίδα. Αυτό το παρατηρούμε και στη χώρα μου και σε άλλες μεσογειακές χώρες. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, στο σημείο 32, όταν μιλάμε για την διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες περιοχές, αλλά και στο εσωτερικό μεταξύ των διαφόρων περιοχών, είναι πολύ σημαντικό της ίδιας χώρας εντός της μίας χώρας γιατί αλλιώς οι λύσεις που θα έχουμε ε, ε, θα είναι λιγότερο αποτελεσματικές και δεν θα δημιουργούν τόσο πολλά απόβλητα. Για την ενέργεια τώρα πρέπει να ευνοήσουμε την αποδοτικότητα και να έχουμε την πρόθεση τεχνολογιών υψηλού επίπεδου αποδοτικότητας και όταν μιλάμε για απόβλητα, μιλάμε για την ανάκτηση και την ανακύκλωση, βεβαίως σωστό, αλλά να αναφέρουμε σαφώς και την ενεργειακή αξιοποίηση των ε, αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών υψηλής απόδοσης. Αυτές τις προσθήκες θα ήθελα στο σχέδιο ψηφίσματος. Ευχαριστώ πολύ. Η... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε εδώ. Ε, οι δυο μας, ε, η Επιτροπή μας και εσείς, ε, τα έχουμε πει επανειλημμένα για το Ρίο για την παγκόσμια συνδιάσκεψη. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μας θέματα. Είναι η θεωρία περί μηδενικών αποβλήτων. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για το τι θέλετε να κάνετε στο Ρίο, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που μας ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και εάν ε, το ε, συνδυάσουμε με αυτά που συζητήσαμε στο Κοινοβούλιο για τις πρώτες ύλες νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πει και αυτή τη γνώμη της. Αυτό είναι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της ε, στρατηγικής ε, φυσικών πόρων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αντικατάστασή τους και αποτελεσματικότητα. Ε, ένα άλλο θέμα το οποίο πολύ συχνά έχουμε συζητήσει είναι η απαγόρευση διατήρησης ε, των αποβλήτων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Οι τιμές ε, των ε, πρώτων υλών αυξάνονται συνεχώς. Παρόλα αυτά όμως εμείς τα πετάμε τα τρόφιμα, τα πετάμε και τα μεταφέρουμε και στον τρίτο κόσμο. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποφύγουμε το dumping. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατάμε, να φυλάμε τα απόβλητα και να προβαίνουμε σε ανακύκλωση. Χαίρομαι που θα γίνει συνάντηση στο Ρίο γιατί εδώ και 20 χρόνια προσπαθούμε το όλο θέμα να το κρατήσουμε στην επικαιρότητα. Δεν πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε αυτή η συνάντηση να είναι απλά μία από τις πολλές για το κλίμα. Δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσουμε ή πρέπει να ξαναμιλήσουμε για ποσοτικά μετρήσιμους στόχους. Αυτό που έχει σημασία είναι να συναντηθούμε, να διαβουλευτούμε και όλοι να ευαισθητοποιηθούμε για το θέμα αυτό, γιατί όπως ε, είπαν και συνάδελφοι, ε, το Globus ε, είναι μια καλή πρωτοβουλία και νομίζω σε αυτό έχει προσχωρήσει το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνάδελφος από το Βελγικό Κοινοβούλιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι στο Βέλγιο, η... στο Μοσουδιακό μας Κοινοβούλιο, η Αρμόδια Επιτροπή ανησυχούσε για το θέμα της πράσινης οικονομίας λέγοντας ότι είναι μια έννοια που αποδυναμώνει τη γενικότερη έννοια της αηφόρου ανάπτυξης. Το παράδειγμα που έδωσε ο κύριος Γερμανάντη και δεν είμαι βέβαιη ότι το παρακολούθησα, αν υποθέσουμε ότι το, η, η, η τώρα ε, εκλείουν λιγότερο διοξίδιο του ε, άνθρακα. Ε, καλό είναι μεν αυτό, αλλά δεν έχουμε λύσει κανένα πρόβλημα σε καμία η οικονομία, ούτε τα ζητήματα δηλαδή της αηφόρου ανάπτυξης, ούτε τα ζητήματα της υποβάθμισης του εδάφους και των δασών. Η πράσινη οικονομία πρέπει να θεωρείται μια ολόκληρη οικονομία η οποία όμως δουλεύει εντό των ορίων ε, της βιοποικιλιότητας ε, της διατήρησης των οικοσυστημάτων, της προστασίας του κλίματος και της χρήσης ε, των φυσικών πόρων. Η, α, η φόρος ανάπτυξης είναι κάτι πολύ ευρύτερο από την πράσινη οικονομία. Οπότε η το θέμα των ε, ε, τιμών νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να αποδυναμώνει τις αρχές αυτές που εδώ και 20 χρόνια ε, θέλουμε να εφαρμόζουμε. Το θέμα της ενέργειας επίσης επιμείναμε εμείς όλος ιδιαίτερος στο Βέλγιο γιατί υπάρχει ιδιαίτερη πίεση όσον αφορά τους, το πετρέλαιο και ε, οι πολλές χώρες πηγαίνουν σε όλο και πιο ευάλωτες ζώνες για να αναζητήσουν πετρέλαιο, σε πιο ευάλωτες χώρες ε, και νομίζω ότι στο Ρίο συν 20 ε, θα έπρεπε να αποθαρρύνουμε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια εξόρυξης πετρελαίου σε οικολογικά ευάλωτες ζώνες όπως για παράδειγμα οι θάλασσες, η Αρκτική ή σε διάφορες περιοχές του Ισημερινού, οι περιοχές που μας ενδιαφέρουν όλος ιδιαίτερος όπως το Κονγκό. Ε, το Βελγικό Κοινοβούλιο είναι υπέρ μιας χρήσης περιορισμένης πυρηνικής ενέργειας και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να αναφερθεί ως τμήμα των ενδεχομένων ε, ε, πηγών, αλλά δεν πρέπει να είναι τμήμα της πράσινης ανάπτυξης. Εμείς θα προτιμούσαμε να μην αναφέρεται ως τμήμα της πράσινης οικονομίας είναι κάτι, κάτι ακόμη επίση ε, που αναφέραμε ε, στο πλαίσιο ε, του Βέλγου απεσταλμένου μας, του κυρίου Ντεσκούτε του ΟΝΟΙΕ, για τα ζητήματα αυτά. Μιλήσαμε για τα θέματα της γεωργίας, της αγροοικολογίας ε, με ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον και του ζητήσαμε να υπερασπιστεί τους γεωργούς και τις πρακτικές που είναι προσβάσιμες ε, ε, από όλους τους μικρούς γεωργούς. Θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το είδος της γεωργίας, όμως αυτό από πλευράς καταναλωτή σημαίνει μία μεταρρύθμιση του διατροφικού συστήματος, οπότε Θυμάμαι τι είπε σε σχέση με αυτό ο Επίτροπος στην αρχή της ομιλίας, τους, ε, της ομιλίας του. Ελπίζω ότι καταλαβαίνουμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν πρέπει να κρύβουμε τις δυσκολίες του τι ακριβώς θα συμπεριλάβει αυτή η πράσινη οικονομία, ούτε να μην καταλαβαίνουμε ακριβώς τι θυσίες θα πρέπει να κάνουν οι χώρες μας. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Λούκας από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Πρόεδρος Με Α, με συγχωρείτε, του, Ισπανικού, του ε- ε- Εστονικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Πρόεδρε, η οικονομική ανάπτυξη έτσι όπως γίνεται τώρα δεν είναι τόσο καλή για το περιβάλλον διότι δεν υπάρχει συνειδητοποίηση της επίπτωσης στο περιβάλλον. Οι πλούσιοι κατασπαταλούν ε, τρόφιμα, την ε, ενέργεια, καταναλώνουμε υπερβολικά. Τα προϊόντα μας, τα προϊόντα που καταναλώνουμε, απαιτούν χρήση τρομερών πρώτων Τι πρέπει να κάνουμε, χρειάζεται ενημέρωση του πληθυσμού, αύξηση της συνειδητοποίησης. Ο Επίτροπος Ποτότσνικ ξέρει πολύ καλά στην προηγούμενη ζωή του εργαζόμασταν μαζί στον τομέα της εκπαίδευσης για χρόνια και νομίζω μπορεί να επιβεβαιώσει το γεγονό ότι η εκπαίδευση, η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ουσιώδης. Για την Εστονία μερικά στοιχεία για τα προγράμματα που μας απασχολούν. Είμαστε σχετικά μικρή χώρα και έχουμε ένα σχέδιο για να αξιοποιούμε, να χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα βάζοντας ε, σημεία φόρτισης σε διάφορα σημεία της χώρας, ούτω ώστε να είναι δυνατή η χρήση του αυτοκινήτου αυτού. Και επίσης έχει πολλά δάση η χώρα μας και μικρή πυκνότητα πληθυσμού. Οπότε έχουμε και πολλά βοσκοτόπια που δεν χρειάζεται να καλλιεργήσουμε Εάν πρέπει λοιπόν να υλοτομηθούν κάποιες περιοχές, έχουμε συστήματα αναδάσωσης, ούτω ώστε τα δάση μας να διατηρηθούν και να επεκταθούν. Στην Εστονία έχουμε επίσης ένα πρόγραμμα εκτεταμένο για το περιβάλλον συνολικότερα και γι' αυτό θα στείλουμε πολλούς εκπροσώπους στην Εστονία. Φυσικά θα χρειαστεί να πάμε αεροπλάνο, δεν μπορούμε να πάμε με εστιοφόρο, αλλά θα συμβάλλουμε ούτως ώστε να αλλάξει ο κόσμος για να είναι πιο θετικός προς το περιβάλλον. Ε, ευχαριστούμε κύριε Λούκας. Και τώρα συνάδελφος του Ρουμάνα Λόμπ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που μας είπατε και το θετικό μήνυμα που εκπέμψατε. Εγώ πάντα θέλω να σκεπτομαι θετικά και νομίζω ότι στο Ρίο πρέπει να αναλάβουμε μια ισχυρή πολιτική δέσμευση έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτό τον ε, χάρτη πορείας ε, πράσινης οικονομίας. Εγώ ε, αγωνίζομαι για την πράσινη οικονομία, γιατί μεσούσεις της κρίσης χρειαζόμαστε περισσότερες λύσεις, χρειαζόμαστε ατμομηχανές για την πράσινη οικονομία. Η πράσινη οικονομία είναι ένα είδος ατμομηχανής είναι σημαντικό να υπάρχουν πράσινες θέσεις εργασίας. Και σας ερωτώ, πιστεύετε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαζόμαστε στρατηγική για την πράσινη οικονομία. Διότι αυτή η πράσινη οικονομία είναι σημαντικό εργαλείο για να επιτύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και το Ρίο πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές ε, είναι άρρηκτα συνεδεμένες μεταξύ τους για να επιτύχουν τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, και την πράσινη ανάπτυξη. Γι' αυτό κάνω αυτή την ερώτηση. Και επιπλέον, διότι εδώ έχουμε και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Οφείλουμε να εκπέμψουμε χειρό μήνυμα προς τις Εθνικές Κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προς την Επιτροπή. Να τους καλέσουμε να μην νοθεύσουν ε, την ε, περιβαλλοντική κοινωνική διάσταση στην πράσινη οικονομία, ακόμα και αν ε, πληττόμεθα από οικονομική κρίση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στο, Ρέο, στο Ρίο με να γίνει μια πραγματική πολιτική συμφωνία και να επιδιώξει αυτό που λέει ο τίτλος της συνάντησης «Το μέλλον που θέλουμε». Επόμενος ομιλητής από τη Δανία, ο κύριος Χάντζεν, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το σύνθημα για το Ρίο είναι 20, το σύνθημα The Future We Want, ε, είναι ένα πολύ καλό σύνθημα. Πολύ καλό σύνθημα και για το μηδενικό σχεδιασμό, διότι αποδεικνύεται ότι εμείς που βρισκόμαστε εδώ και οι συνάδελφοί μας, εμείς είμαστε εκείνοι που μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία, ε, να λάβουμε τις σωστές πολιτικές αποφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό τα Εθνικά Κοινοβούλια και οι κοινοτικοί θεσμοί να έχουν κατά νου ότι στο Ρίο δεν θα δρομολογηθούν νέες διαδικασίες. Απλά θα υπάρξουν δεσμευτικοί στόχοι γιατί αλλιώς ε, μετά από κάποια χρόνια απλά θα διαπιστώσουμε ότι δεν προχωρήσαμε. Το Ρίο είναι μια περιβαλλοντική συνδιάσκεψη η οποία θα ασχοληθεί ε, με στόχους ε, βιωσιμότητας θα ασχοληθεί με την κοινωνική βιωσιμότητα ε, και την περιβαλλοντική. Ε, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι τομείς της ε, πολιτικής. Έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες για να επιτύχουμε όλα αυτά, αλλά θα αντιμετωπίσουμε και προβλήματα. Έχουμε πολλές γνώσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα του πλανήτη, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έγιναν πάρα πολλά και αυτό είναι παράδοξο το κέρδος ε, υπολογίζεται μακροπρόθεσμα, ε, όμως το εθνικό κέρδος υπολογίζεται βράχυπρόθεσμα. Άρα δηλαδή εμείς, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Κοινοβούλια οφείλουμε να επιδιώξουμε δεσμευτικούς στόχους. Οφείλουμε να συνεχιστούν οι να μεριμνήσουμε για να συνεχιστούν οι πολιτικές διαδικασίες. Ε, καθαρό νερό, ε, βιώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικοί ε, στόχοι. Αλλά δεν πρέπει όλα αυτά να τα μεταθέτουμε στις ελληνικές ε, καλένδες. Και κάτι άλλο. Θα πρέπει να καταβληθεί ένα τίμημα και επανέλθουμε στον Sir Humber Storms, ο οποίος το 2006 συνέταξε μια έκθεση και είπε ότι το τίμημα της αδράνειας είναι πολύ ψηλότερο από το τίμημα της πράξης, της δράσης. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε κατά νου. Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τίμημα της αδράνειας θα είναι σημαντικότερο από το να καθορίσουμε δεσμευτικούς στόχους ε, στις ε, προτεραιότητές μας. Ε, the future we want, αυτό το ορίζουμε μόνοι μας και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Συνάδελφος Νίγκρι από το Λουξεμβούργο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτρόπε, έχετε δίκιο που μιλάτε για κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως θα ήθελα μία ακόμη φορά να θέσω πάλι το θέμα της θέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, σε σχέση με τις χώρες που δεν συμμετείχαν ε, στο πρωτόκολλο του Κιώτο. Έχουμε τη στρατηγική τρεις φορές 20 για το 2020 με όλους σχετικούς μηχανισμούς. Νομίζω ότι το Ρίο θα έπρεπε να συμπεριλάβει όλο τον κόσμο και κάτι ακόμη που θα ήθελα να θέσω. Είπατε ότι μεταξύ των πρώτων στόχων είναι οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, κάτι το οποίο μου οδηγεί σε δύο ερωτήσει. Το πρώτο ερώτημα αφορά τα αγροπεριβαλλοντικά ε, προϊόντα, όπω επίση και την παραγωγή βιοκαυσίμων. Ε, αυτά όλα συνάδουν με την νέα ε, γεωργική πολιτική την γεωργική πολιτική του 2013 ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να, να, να θρέψουμε 9 δισεκατομμύρια στόματα και Μία ακόμη ερώτηση για τις χώρες που λαμβάνουν αναπτυξιακή βοήθεια. Μήπως μπορούμε να τους ενθαρρύνουμε για τη χρήση ε, της ηλιακής ενέργειας ε, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα της ΕΡΤΑΚ για παράδειγμα. Ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στην Αφρική. Θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε περισσότερο την ηλιακή ε, ενέργεια, κάτι που γίνεται λιγότερο στις χώρες της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ρίχα Ευχαριστώ. Είπατε πολλά για την πράσινη οικονομία. Ξέρουμε ότι αν δεν την επιτύχουμε, μακροπρόθεσμα στον πλανήτη, στον πλανήτη θα έχουμε ένα πρόβλημα ως ε, άνθρωποι. Αλλά το θέμα είναι ε, αυτά που μας προσφέρουν τα οικοσυστήματα να τους δώσουμε μια συγκεκριμένη τιμή, να τους αποδώσουμε. Είστε οικονομολόγος αρχικά. Καταλαβαίνετε ότι συχνά στην οικονομία χρειαζόμαστε τιμές για να εργαστούμε. Πολλά λοιπόν από αυτά τα πράσινα προγράμματα τα διάφορα, για παράδειγμα, διάφορες καταστάσεις ε, παραγωγής ενέργειας θέλουν επιδοτήσεις. Αν δεν μπορέσουμε να έχουμε σωστές τιμές, δηλαδή αυτό το εξωτερικό κόστος να ενταχθεί στο κόστος παραγωγής, δεν θα λειτουργήσουν αυτές οι καταστάσεις. Και έχω ανησυχίες. Πόσο δύσκολο ήταν, για παράδειγμα, προσπαθώντας να περιληφθεί στον τομέα των μεταφορών το κόστος αυτό στον υπολογισμό του κόστους. Χρειαστήκαμε περίπου 20 χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι να φτάσουμε σε κάποιους κανονισμούς που ε, οριακά είναι ικανοποιητικός. Αύριο θα μιλήσετε για θέματα νερού. Αλλά κύριε Επίτροπε έχουμε το περίφημο άρθρο 9 θα μας κάνετε πρόταση για κατευθύνες γραμμές για το πώς θα μπορέσουμε να επανακτήσουμε το κόστος. Υπάρχουν πολύ διαφορετικά συστήματα στα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει σαφής κατεύθυνση. Πώς θα κανονίσουμε την τιμολόγηση των υδάτων σε κάθε χώρα. Γιατί είναι διαφορετικά τα συστήματα. Να έχουμε σωστές τιμές, γιατί αλλιώς σε μικρό επίπεδο δεν μπορεί να υπάρξει κανονισμός αλλά συνολικά η κοινωνία σε μακροοικονομικό επίπεδο πρέπει να φέρει το κόστος. Ευχαριστώ, Ρίχαρτ. Ο συνάδελφος Μπάσλε από το Σλοβενικό Κοινοβούλιο. Χαίρετε, κύριε Επίτροπε, που είστε από την ε, Σλοβενία. Συγχαίρω τους, συναδέλφους που μπορούν μετά από ένα τόσο καλό μεσημεριανό φαγητό συνεχίζουν να μπορούν να ε, συζητήσουν τόσο σωστά. Γιατί όπως ξέρετε μετά από ένα τέτοιο φαγητό η ιατρική λέει ότι πρέπει να κάνει, πάρει κανείς έναν υπνάκο. Αλλά παρόλα αυτά μια χαρά συζητήσεις κάνουμε. Η Σλοβενία υποστηρίζει τη διοργάνωση Ρίο Συνήκωση. Χαιρόμαστε πολύ που υπάρχουν τόσο υψηλές προσδοκίες ότι θέλουμε να καθορίσουμε δεσμευτικούς στόχους που να βοηθήσουν την περαιτέρω επίτευξη της πράσινης ανάπτυξης, την εξάλληψη της ε, φτώχειας επίσης. Η Σλοβενία ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη των θεσμικών οργάνων. Για την ε, Σλοβενία είναι σημαντικό να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον και την περιβαλλοντική διάσταση η διάσκεψη Ρίο συν θα έπρεπε να καλύψει και τους τρεις τομείς, τον οικονομικό, κοινωνικό και οικολογικό. Η Σλοβενία παίζει ενεργό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, οι προσπάθειες αυτές. Έχουν γίνει από τη Σλοβενία εδώ και πολύ καιρό. Το πρωί ακούσαμε πολύ αισιόδοξε τοποθετήσεις, ίσως υπερβολικά αισιόδοξε, σαν να είχαμε όλοι ήδη αποφασίσει δεσμευτικούς στόχους. Έχω όμως την αίσθηση, κύριε Επίτροπε Ποτότσνικ, είπατε και εσείς στην ομιλία σας ε, ότι έχετε κάποιες επιφυλάξεις, ε, κάποιο σκεπτικισμό για την ε, πολιτική βούληση άλλου να συνεργαστούν μαζί μας αυτή τη συνέλευση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άχερτ. Ο Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον Επίτροπο, αλλά έχω και μία συγκεκριμένη ερώτηση. Δηλαδή, μετά τον Ντόρμπαν, ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που συνέβη στον Ντόρμπαν ήταν η συμμαχία ανάμεσα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και τις περίφημες low-lying countries. Τι πιστεύετε εσείς, ε, πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η συμμαχία. Ε, είναι σημαντικό το Στορίο να προχωρήσει αυτή η συμμαχία με τις ανεψόμενες χώρες και τις χώρες με χαμηλό υψόμετρο. Αυτό που επίσης είναι καθοριστική σημασία στο Ρίο δεν είναι μόνο να μιλήσουμε για την πράσινη οικονομία αλλά και για αυτές τις συμμαχίες. Μήπως μπορείτε λοιπόν να μας διευκρινίσετε ακριβώς ε, ε, τι πιστεύετε από αυτού. Και κάτι άλλο που θέλω να πω σε όλους σας. Πάρα πολύ ωραία να μιλάει κανείς για την ε, πράσινη οικονομία. Ε, όλοι συμφωνούν πόσο σημαντική είναι, αλλά παράλληλα όλοι γνωρίζουμε ότι η πράσινη οικονομία ξεκινάει στην πατρίδα μας. Και ένα από τα πιο απλά πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε είναι να αλλάξουμε τη φορολογία. Να επιβάλλουμε φόρο στην οικολογική επιβάρυνση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόταση για ενεργειακό φόρο. Να περάσουμε από τον όγκο σε περιεχόμενο ε, διοξιδίου και περιεχόμενο ενέργειας. Είναι απλά μετατόπιση των κανονισμών. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό να γίνει, αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι στην Ευρώπη, όταν πρόκειται για φορολογικά θέματα, ε, τα κράτη-μέλη, το καθένα από αυτά ε, καταθέτουν βέτο. Μία χώρα μπορεί να μπλοκάρει, ε, ας πούμε, το Λουξεμβούργο. Και στρέφομαι στους αδέλφου ε, από το Λουξεμβούργο που μιλάνε για την πράσινη οικονομία. Ένα, ορίστε, ειδού η ευκαιρία να αλλάξετε τη φορολογία σας, να αντιμετωπίσετε το περιβαλλοντικό βάρος, Κατανοώ ότι θέλετε εδώ να μας στηρίξετε, αλλά πρέπει να κάνετε ορισμένα απλά πράγματα. Γιατί όταν θέλετε να μιλάτε για την πράσινη οικονομία, να αλλάξετε τη φορολογία. Και αυτό να το κάνουν και τα 27 κρατημέλη, για τελειώ απλά χάνουμε το χρόνο μας και τίποτα δεν θα γίνει ιστορίο. Και λυπάμαι, θα ήταν κρίμα να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Άιχορτ. Τελείωσε ο κατάλογος ε, των ερωτώντων και τώρα θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στον Επίτροπο να απαντήσει γιατί ετέθησαν ορισμένα θέματα ε, και μπορεί ο Επίτροπος να κάνει και μια γενικότερη ε, ανακεφαλαίωση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή συζήτηση αυτή που έγινε και θα ήθελα να τοποθετηθώ σε όλες τις ερωτήσεις, σε μερικές θα είμαι πιο σύντομο, σε άλλες θα ε, αφιερώσω περισσότερο χρόνο για να σας εξηγήσω λιγάκι το σκεπτικό μας. Πρώτα απ' όλα, ε, απευθύνομαι στον ε, συνάλφα από την Μάλτα. Πράγματι, οι δείκτες εντάσσονται μέσα στο σκεπτικό μας. Σωστό αυτό που είπατε. Δεν είναι ότι όλα ταιριάζουν για όλους. Αυτό θα ληφθεί υπόψη. Τώρα, Όσον αφορά τη διασύνδεση. Κοιτάξτε, έχουμε τους στόχους της χιλιετίας και έχουμε και κάτι που αυτή τη στιγμή περίπτεται ως μήνυμα. Ένα λοιπόν από τα μηνύματα που κυκλοφορούν είναι ότι στο Ρίο πρέπει να συμφωνήσουμε για τη δρομολόγηση της διαδικασίας που θα οδηγήσει προς την βιωσιμότητα. Δύσκολο βέβαια να πει κανείς όχι σε αυτό, αλλά εμείς ως Ευρωπαίοι αυτό που προσθέτουμε είναι το εξής. Αν θέλουμε η διαδικασία αυτή να είναι αξιόπιστη, τότε είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε καθαρές συμφωνίες στο Ρίο. Η αλλιώ ε, θα καταλήξουμε σε πολιτικές δηλώσει που δεν θα είναι όμως δεσμευτικές και δεν θα κατησυχάζουν τους πολίτες ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Άρα δηλαδή αν θέλουμε να στηρίξουμε την έννοια των, των SDGs, ε, αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε και μέσα από τους ε, στόχους μας. Να δούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τους δικούς μας τους στόχους. Να δώσουμε λοιπόν μια αξιοπιστία στις δραστηριότητες μας σε σχέση και με τους, ε, το μέλλον. Το τρίτο θέμα ε, και εδώ νομίζω πρέπει να σταθώ περισσότερο. Κοιτάξτε, Ας δούμε τον αναπτυσσόμενο κόσμο και τι κάνουμε σε αυτή τη μεταβατική φάση. Πρώτα απ' όλα, αν δούμε το θέμα από το πρίσμα του πού ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, θα διαπιστώσουμε ότι η άποψη ότι θα προσκρούσουμε σε τείχο λόγω του ότι είναι πεπερασμένοι η φυσικοί πόροι, αυτό Νομίζω ότι είναι σαφές. Εκείνο για το οποίο προσπαθούμε να πείσουμε τους άλλους είναι ότι και οι χώρες εκείνες οι οποίες ε, μοιάζουν να έχουν περισσότερους πόρους και λιγότερους περιορισμού, κατ' ουσίαν βρίσκονται ε, στο ίδιο πλοίο, στην ίδια μπάρκα. Ίσως ε, να έχουν ακόμα κάποιες ευκαιρίες που δεν έχουμε εμείς, ίσως αυτοί να μπορούν να αποφύγουν την επώδυνη μεταβατική διαδικασία για την οποία μιλήσατε πολύ. Βεβαίως ε, επικαλούνται ε, τα μοντέλα παραγωγή ε, και κατανάλωση και ξέρετε ότι η συνήθεια των ανθρώπων είναι το τελευταίο και πιο δύσκολο πράγμα να αλλάξει. Κατά κάποιον τρόπο, εμεί είμαστε περισσότερο αναγκασμένοι από του άλλου να αλλάξουμε. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμά μα. Αν όλοι προσπαθήσουμε από κοινού, τότε ενδεχομένω να αποφύγουμε κάποια λάθη ε, σαν αυτά που έγιναν από κάποιους και τα βλέπουν οι άλλοι που έχουν λιγότερους πόρους. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι σαφέ σαφές μήνυμα. Ότι κατ' ουσίαν όλοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να γίνει κατανοητό ότι όταν μιλάμε για την πράσινη οικονομία, μιλάμε κατ' ουσίαν για το ίδιο πρόβλημα για όλου. Ίσως κάποιοι να το κατανοούν καλύτερα από του υπόλοιπου και άκουσα κάποιου να λένε ότι αυτό συνδέεται με την κρίση που μαστίζει την Ευρώπη. Κοιτάξτε, συνδέεται με την Ευρώπη με την έννοια ότι ε, η ιδέα αυτή επικρατεί, αλλά έχουμε συζητήσει για τέτοιου είδου θέματα και πριν από την κρίση. Αν θέλετε όμω οπωσδήποτε το θέμα αυτό να το συνδέσετε με την κρίση, υπάρχουν αποχρόντε λόγοι που οδηγούν στο ότι πολύ εύκολα συνδέεται το θέμα αυτό με την κρίση. Ε, αν θέλετε ε, να συνδέσει το θέμα με, την, ε, με τα χρέη που έχουν αληφθεί, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη και για να υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη πρέπει κανεί να είναι περισσότερο ανταγωνιστικό. Και πού θα τη βρει αυτή τη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αυτά λοιπόν τα μαγικά συσταγωγικά θέματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη γιατί πραγματικά ε, έχουμε πρόβλημα με την ανταγωνιστικότητα. Η οικονομία τη γνώση εδώ είναι σαφέ. Αν έχουμε καλά εκπαιδευτικά συστήματα, ερευνητικά, ε, καινοτόμα συστήματα, πολύ ωραία. Όμω, κάτι ε, το οποίο επιδιώκουμε και το επιδιώκουν και οι επιχειρήσεις, ε, όπως είπε και ο κύριος Γκεμπράντη, υπάρχει αυτό που ψάχνουν και οι επιχειρήσεις έχουν κατανοήσει πολύ καλά ότι αν δεν παράγουν τα προϊόντα χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια, νερό, υλικά, να τα παράγουν με ένα τέτοιο τρόπο να μπορούν να ανακυκλώνται, τότε και οι αγορέ ε, οι επιχειρήσεις αυτές θα εξαφανιστούν από την αγορά. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει κατανοητό. Γι' αυτό οι επιχειρήσεις πάνε από την παραγωγικότητα της εργασίας στο παρελθόν, όπου η πόλη ήταν φτηνή και το κόστος εργασίας πολύ ψηλό και έτσι έφτιαξαν κάποια συστήματα παραγωγής ε, όπου δεν χρειαζόντουσαν πλέον την ανθρώπινη εργασία. Δεν είναι όμως δυνατόν να παράγει κανείς χωρίς φυσικούς πόρους. Ε, στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, σήμερα το 45% στο κόστος ε, μιας ε, εταιρείας είναι οι πόροι και το 20% είναι μόνο το κόστος ε, της μισθοδοσίας. Άρα δηλαδή, αν θέλει κανείς να σκέφτεται περιβαλλοντικά, πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτό που υπάρχει και δεν πρέπει να εξαφανιστεί. Άκουσα κάτι για την πράσινη ανάπτυξη. Ε, ότι αυτή είναι η έννοια που χρησιμοποιεί ο αναπτυγμένος κόσμος για να αναχαιτήσει το μοντέλο ανάπτυξης. Κοιτάξτε, δεν θα μιλάγαμε για την πράσινη ανάπτυξη αν υπήρχε κάποιο λάθος με την καφέ, όπως τη λέμε, ανάπτυξη. Δεν θα την αναφέραμε καν, διότι η απάντηση, μάλλον η πράσινη ανάπτυξη έχετε δικά της τα όρια και η πράσινη ανάπτυξη είναι η απάντηση σε αυτό πώς δηλαδή μπορούν να ληφθούν ορισμένα πράγματα υπόψη που αγνοήσαμε κατά το παρελθόν όταν είχαμε παραγωγή και πώς μπορούμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη γιατί αλλιώ θα προσκρούσουμε σε τείχο. Αυτό νομίζω ότι είναι προφανές. Ο ιδιωτικό τομέα τώρα κάτι που το αναφέρατε πολύ από εσά. Όταν μιλάμε για την πράσινη οικονομία και ανάπτυξη, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να μιλάμε αγνοώντας τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, όταν μιλάμε για μέσα εφαρμογής. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για μέσα εφαρμογής εδώ, είναι διαφορετικό αυτό από αυτό που αναφέρεται πολλές φορές στο πλαίσιο της ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Γιατί, διότι αν θέλει κανείς να φτιάξει ένα πραγματικό μοντέλο πράσινης ανάπτυξης, το σημαντικότερο είναι να δημιουργήσει κανείς τις συνθήκες, μέτρα στην αγορά, συνθήκες οι οποίες προσελκύουν τους επενδυτές αυτούς τους τομείς. Και βεβαίω ε, χρειάζεται κανεί και την δημόσια, την κρατική υποστήριξη. Αλλά δεν γίνεται όμως αυτό να επιτευχθεί μόνο με τη μεταφορά κονδυλίων διασυνοριακά, αν κάποιο ε, δεν ε, αλλάζει προ τη κατεύθυνση μόνο του στην πατρίδα του, αυτό δεν βοηθάει. Και όσον αφορά την εξάλληψη της φτώχειας, είμαι ακράδαντα πεπισμένο ότι η εξάλληψη της φτώχεια δίνει τη δυνατότητα στου ανθρώπου να ζουν διαφορετικά. Η δημοκρατία, Του δίνει τη δυνατότητα να ζουν σε δημοκρατία, να έχουν υπηρεσίε υγεία, παιδεία, όμως τους δίνει επίσης τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο νερό, ε, πρόσβαση στην ενέργεια και σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη διατήρηση των οικοσυστημάτων. Το να καταστρέψει λοιπόν κανείς αυτά τα οικοσυστήματα κατ' ουσίαν τι σημαίνει τους εξωθεί κανείς τη φτώχεια. Και νομίζω το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι πολύ καλά αυτό. Και όλοι μας ε, πρέπει να αγωνιστούμε να μην στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, γιατί μιλάμε για αυτούς τους ε, πέντε τομείς ε, που σας παρουσίασα. Ίσως λιγάκι πρέπει να σας το εξηγήσω καλύτερα για να το καταλάβετε. Υπάρχει τώρα πλημμυρίδα ιδεών που κυκλοφορούν και αν δεν εστιάσει κανείς την προσοχή του σε ορισμένα πράγματα που θα βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας, τότε δεν θα μπορέσουμε να έχουμε σαφή προσέγγιση και συστηματικοποίηση της σκέψης στην Ευρώπη. Όπως είπα και προηγουμένως, το καλύτερο απ' όλα είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας στον καθορισμό στόχων σε κάποιους τομείς που όπως σας είπα προηγουμένως αποκαλούμε πυλώνες ζωής. Πρώτον, ε, βιώσιμη ανάπτυξη, κάτι που το είχε ε, προτείνει και ο Μπανκιμούν και το βιώσιμο πάνελ. Αυτό ε, είναι το καλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεύτερο, νερό. Ήδη έχουμε τους στόχους της χιλιετίας που μιλάνε για το ε, νερό για όλους, ε, για την υγιεινή. Ε, σημαντική λοιπόν είναι η επάρκεια. Η επάρκεια νερού είναι καθοριστική σημασία για χώρες που είναι στην κατώτατη στάθμη της ανάπτυξης που χρησιμοποιούν όλα τα αποθέματα για τη γεωργία. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό, οι χώρες αυτές θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα ανάπτυξης και εξάλληψης της στόχιας. Κατόπιν, διαχείριση της γης, ε, το να αναχαιτήσουμε την επιδείνωση των οικοσυστημάτων. Αυτό είναι το σημαντικότερο για τις ε, χώρες της Αφρικής. Όταν μιλάμε για τους ωκεανούς και για τα ενάλια οικοσυστήματα, Κοιτάξτε, οι ωκεανοί είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας. Από την άλλη όμως είναι και καθοριστική σημασίας ε, και για τους πλέον, για ένα από τα ευάλωτα νησιά στον Ειρηνικό. Και όταν μιλάμε για το πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πυλώνες οι οποίοι είναι το συστατικό, θα αποτελέσουν στο μέλλον το συστατικό της ζωής μας, Βεβαίω και οι βιώσιμε πόλει είναι σημαντικέ. Αν όμω δεν αντιμετωπίσει κανεί το νερό, την ενέργεια, τα απόβλητα, μπορεί κανεί να ξεχάσει τι βιώσιμε πόλει. Ή, παραδείγματο χάρη, η επισητιστική ασφάλεια που είναι και αυτή είναι πολύ σημαντική. Μα φυσικά δεν τα αμφισβητεί κανεί. Όμω μακροπρόθεσμα αυτή μπορεί κανεί ε, να αντιμετωπίσει μόνο μέσα από την αναχέτηση τη επιδείνωση των οικοσυστημάτων και με την καλύτερη χρήση του νερού. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτά είναι εργαλεία δράση που μπορούν να υπάρχουν στο χάρτη πορείας και θα πρέπει να ακολουθήσει κανείς ε, κάποιες ε, από αυτές ε, τις φέρουσες κολόνες του σπιτιού προσπαθούμε να χτίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας στους πόρους. Όχι να αναμειγνύουμε το θέμα αυτό με τους τομείς ή με λειτουργικές δραστηριότητες. Ωραία όλα αυτά, είναι κάτι που κανείς μπορεί να τα εξηγήσει και να αποκτήσουν και νόημα. Η κυρία Μέρκης, μη συγχωρείτε, απαντώντας στην κυρία Μέρκης, μας ε, ζήτησε το Συμβούλιο να ασχοληθούμε με τους στόχους και ασχολούμαστε με τους στόχους και με τα απόβλητα που μπορεί να προταθεί και για το Ρίο πολύ ελκυστικό είναι για παράδειγμα τα τροφικά απόβλητα που δεν αφορά μόνο τις ε, αναπτυγμένες αλλά και τις αναπτυσσόμενες χώρες για πολύ διαφορετικούς λόγους. Αλλά εάν κάποιος θεωρεί ότι δεν μπορούμε να θρέψουμε τα 9 δις που θα έχουμε το 2050 με ό,τι παράγουμε τώρα, μπορούμε με ό,τι παράγουμε τώρα. Γιατί σπαταλούμε τόσα τρόφιμα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Και πολλά άλλα αναφέρατε για τις ε, χωματερές ε, και νομίζω ότι η φορολόγηση των ε, χωματερών θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσουν οι χωματερές, αλλά είναι δύσκολο να το επιβάλλουμε σε κάποιες χώρες. Αν συμφωνήσουμε για τις πολιτικές σε αυτό το τομέα, επειδή εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι στο κέντρο της προσοχής τα απόβλητα στο Ρίο, μπορούμε να επιτύχουμε ορισμένα πράγματα. Βεβαίως, η εκπαίδευση για το περιβάλλον. Συμφωνώ απόλυτα. Κάτι άλλο, σύντομα. Η πράσινη οικονομία. Και ποια είναι η προσέγγιση μας. Ρωτήσατε εάν την έχουμε. Βεβαίως, βεβαίως, η αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων είναι το μάντρα μας. Ίσως δεν ε, συμπεριλαμβάνουμε όσο πρέπει την κοινωνική πλευρά. Αλλά όλα αυτά τα συστατικά είναι τμήμα της προσέγγισης μας. Αν θέλουμε να επιτύχουμε την πράσινη οικονομία, να καταλάβουμε τα εξής. Δεν υπάρχει πανάκια. Χρειάζεστε μέτρα για την αγορά. Χρειάζεστε κανόνες, νομοθεσία. Χρειάζεστε πρόθεση, χρειάζεται καλή έρευνα και ανάπτυξη, δημόσια στήριξη. Όλα αυτά χρειάζονται. Άρα χρειάζεται μια πολιτική προοπτική και πολιτική αποφασιστικότητα. Χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν γίνεται τίποτα. Και χρειαζόμαστε και εταιρικέ σχέσεις, δημόσιες, ιδιωτικές, διασυνοριακές. Κάτι λοιπόν σαν αυτό που λέμε ότι θέλουμε να επιτύχουμε στο Ρίο. Ναι, είμαστε υπέρ δεσμευτικών στόχων. Έχουμε τα πορίσματα του Συμβουλίου, γι' αυτό, για τη σχέση με το Κιώτο. Βεβαίως, να εργαστούμε με βάση τη συμφωνία του Ντέρμπαν, με μεγάλη συμμετοχή των Ευρωπαίων αποφασίστηκε βιοκαύσιμα. Η άμεση απάντησή μου είναι κριτήρια βιωσιμότητας. Ό,τι πολιτική δημιουργείται δεν θα πρέπει να δίνετε κάτι με το δεξί, να το παίρνετε με το αριστερό. Η βιωσιμότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ευρύτερη έννοια. Απόλυτα ισχύει και για τα βιοκαύσιμα αυτό. Ανάπτυξη στην Αφρική. Είπα τις συνθήκες που θα βοηθήσουν να υπάρξει. Μέτρα για την αγορά βεβαίως. Τέλος. Για αυτήν τη συμμαχία και τον σκεπτικισμό που ανέφερε ο συνάδελφος από τη Σλοβενία. Μην νομίζετε ότι συμφωνούν όλοι με τα μέτρα τα οποία προτείνουμε. Είναι τεράστιο ενώπιόν μας για να τους πείσουμε όλους ότι είμαστε ειλικρινεί σε αυτά που κάνουμε και ότι μπορεί να βασιστούν σε μας. Δεν πρόκειται για προσπάθεια προστατευτισμού, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τίποτα στους άλλους, αλλά ίσως λόγω των συνθήκων ζωής μας ορισμένα θέματα τα καταλαβαίνουμε καλύτερα από άλλους. Η πραγματικότητα όμως αποδεικνύει ότι όλοι είμαστε στην ίδια βάρκα. Αν νομίζουν ότι μπορούν να συνεχίσουν το πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης το σημερινό, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα και στο μέλλον. Να το καταλάβουμε λοιπόν αυτό. Η φιλοδοξία μας θα αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Όπου θα πρέπει να είμαστε πιστικοί. Σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 4,5 ώρα στη Βραζιλία πίστηκα ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Γιατί η Βραζιλία δεν είναι χώρα όπου βλέπουν ότι οι πόροι φτάνουν στα όρια τους. Έχει πολλούς πόρους η χώρα. Αλλά καταλαβαίνουν πολύ σοβαρά τα περιβαλλοντικά θέματα. Υπάρχει περιβαλλοντικό κίνημα, σε όλες τις χώρες υπάρχει, ούτως ή άλλως. Να καταλάβουμε όμως ότι δεν ισχύει ότι όλοι καταλαβαίνουμε τον ίδιο τρόπο τα προβλήματα και τις λύσεις. Αναφερθήκατε σε συμμαχίες. Βεβαίως πρέπει να τις επιτύχουμε. Αξίζει τον κόπο να εργαστούμε για τη συμμαχία με, τις, ε, με τα μικρά νησιά, με τις αφρικανικές χώρες. Αυτό δεν έγινε μόνο στον Τέρμπαν και στον Αγκόγια έγινε. Στον Durban ίσως ήταν πιο προφανές. Αλλά τώρα είναι ορατό. Είναι απτό. Πρέπει να το προωθήσουμε. Θα έχουμε μια διάσκεψη στην Στοκχόλμη τον Απρίλιο. Άλλη μια καλή ευκαιρία νομίζω. Αλλά δεν θα χάσουμε καμιά ευκαιρία Πολλές θα μπορούσα να αναφέρω για να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε αυτές τις συμμαχίες. Το έχουμε κατά νου. στα πλαίσια της πορείας προς το Ρίο και για το δίκτυο Globe. Καλή ιδέα. Χθες συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βραζιλίας. Μου είπε ποιοι είναι οι στόχοι τους μου είπε πώς προτίθενται να συνεχίσουν να εργάζονται. Δεν είναι δικό μου θέμα τώρα να σχολιάσω, γιατί είμαι από την άλλη πλευρά, αλλά είναι καλή ιδέα. Αξίζει να επενδύσουμε σε αυτήν. Ευχαριστώ Γιάννος Πουτόσνικ που συμμετείχατε, που απαντήσατε σε ερωτήσεις. Για άλλη μια φορά εντυπωσιακά διαπιστώσαμε ότι έχετε σοβαρά την πρόθεση να κάνετε κάθε προσπάθεια να αναφέρετε σωστά επιχειρήματα για να επιτύχει το Ρίο αλλά ότι δεν θα είναι βόλτα στο πάρκο. Δεν θα είναι απλό. Το διαπιστώνουμε και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και εσείς συνάδελφοι στα Εθνικά Κοινοβούλια όταν μιλάει κανείς για βιώσιμη ανάπτυξη με συγκεκριμένες προτάσεις ή με πολιτική κλίματος, τότε η εφαρμογή είναι πάντα δυσχερής, ιδιαίτερα δυσχερής. Αλλά είμαι σαφώς πεπισμένος ότι μπορούμε να σημειώσουμε επιτυχίες. Έχουμε τρεις μήνες καιρό και νομίζω ότι ήταν μια καλή αρχή η σημερινή μας συνάντηση, ούτως ώστε και στα κράτη-μέλη να ξεκινήσει μια συζήτηση για το τι θα επιδιώξουμε τον Ιούνιο στο Ρίο. Για να επηρεάσουμε την πορεία του πλανήτη. Εάν συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα, θα μας ε, κοστίσει πολλά χρήματα. Νομίζω πως και σήμερα αναφέρθηκε και εξηγήθηκε σαφώς. Μιλήσανε για τη συμπερίληψη όλων των στοιχείων κόστους. Χρειαζόμαστε μια έντιμη συζήτηση για το θέμα αυτό. Είναι σαφές Είναι σαφές λοιπόν ότι κοστίζει χρήματα η μετατροπή της οικονομίας μας σε βιώσιμη οικονομία. Σήμερα το πρωί το συζητήσαμε, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, ούτω ώστε τα θεσμικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών να αναδομηθούν. Νομίζω ότι σε πολλές συναντήσεις ε, κατέστη σαφές ότι δεν είναι η καταλληλότερη η τωρινή τους δομή Περιμένω λοιπόν να δω αν θα καταφέρουμε να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια αναδιάρθρωσης στο Ρίο και η ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, η βιώσιμη παροχή ενέργειας και γενικότερα η ενεργειακή αποδοτικότητα μπορούν να συνδυαστούν και αν θα επιτύχουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Εθνικά Κοινοβούλια να υιοθετήσουμε και τα κατάλληλα νομοθετήματα, δηλαδή δεσμευτικές συμφωνίες σημαίνει ότι πρέπει κατόπιν να έχουμε και δεσμευτικά νομοθετήματα. Και όπως είπα δεν είναι πάντα απλό αυτό. Σήμερα διαπίστωσα ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη απόκληση αλλά, το ότι, αλλά και επικάλυψη, αλλά και ότι σε άλλους τομείς πρέπει να επιδιώξουμε να ενδιαφερθούν για, την συνάντηση, για τη συζήτηση αυτή και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με άλλους τομείς. Βεβαίως έχουμε οικονομική κρίση, τώρα η οικονομική κρίση προκάλεσε κρίση χρέους και διάφορα άλλα τμήματα του κόσμου εξετάζουν γιατί η Ευρώπη είναι σε κρίση και πώς θα καταφέρει να ξεπεράσει την κρίση. Πιστεύω ότι η βιώσιμη οικονομία μπορεί να συμβάλλει στην ε, υπέρβαση της κρίσης και έτσι να δώσουμε σημαντική συμβολή στο πώς θα μπορέσουμε να θρέψουμε ένα πλανήτη με 9 δισεκατομμύρια το 2050, ούτως ώστε το 2050 η ζήτηση ενέργειας να μην ανέβει επί τρία από ό,τι σήμερα. Γιατί τότε θα έχουμε μια τεράστια πρόκληση. Πρέπει να συνδυάσουμε περιβάλλον, κλίμα, ανάπτυξη και οικονομία. Και αυτή θα είναι η διαλύθωση συνολικά για την Ένωση, εάν θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτήν την κρίση. Γιατί έχουμε ένα ε, εγγενές ελάττωμα η φορολογική πολιτική, η δημοσιονομική πολιτική δεν είναι κοινοτική αρμοδιότητα, αλλά εθνική αρμοδιότητα. Και οι Υπουργοί Οικονομικών θέλουν να διατηρήσουν φυσικά αυτή την εθνική αρμοδιότητα. Αλλά εάν δεν υπάρξει, για παράδειγμα, φόρος για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, τότε δεν θα έχουμε και επαρκή φορολογικά έσοδα. Είναι ένα μεγάλο εγγενές ελάττωμα αυτό, ίσως είναι λιγάκι προκλητικό αυτό που λέω, αλλά δεν το λέω τυχαία. Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό το θέμα. Τι όργανα δηλαδή, όχι μόνο στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά τι όργανα και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσουμε για να υπάρξει βιώσιμη οικονομική πολιτική. Σας ευχαριστώ θερμότατα, αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, που ε, κάνατε αυτό το μακρύ ταξίδι για να έρθετε στις Βρυξέλλες σήμερα. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή και οι προτάσεις σας από τις διάφορες χώρες μέλη. Τη θεωρώ απλώς μία αρχή. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Καλή επιστροφή. Και ελπίζω στη συνδιάσκεψη του Ρίο που θα είμαστε μόνο 27 από τις 149 χώρες να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες συμμαχίες για έναν καλύτερο κόσμο, όπως το είπε και ο κύριος Επίτροπος. Περί αυτού πρόκειται, τίποτα περισσότερο αλλά και τίποτα λιγότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με τη συνεδρίασή μας και έχουμε μπροστά μας ε, δύο ακόμα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα με το 15, σημείο υπερθμών 15 της ε, ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την πολυανθεκτική φυματίωση στην Ευρώπη. Και εδώ θα συζητήσουμε με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων, ή e CDC όπως λέγεται ε, ως ακρονίμιο, όπως χρησιμοποιείται, και χαιρετίζω κοντά μας και εκπροσώπους του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο κύριος Ρομπέρτο Ρομπερλίνη θα μιλήσει εκ μέρους ε, του ΠΟΗ και επίση έχουμε και τον κύριο Σπρέγκα εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων. Άδειε από ό,τι βλέπω η αίθουσα. Ich möchte dann als erstes Herrn Bertolini das Wort geben für die... Λοιπόν, δίνω το λόγο στον κύριο Μπερτολίνη, αλλά μισό λεπτό, ο, κύριο κύριος Λίζα θέλει το λόγο. Κοιτάξτε, ε, η Έστερ Λάγκε ζήτησε να μπει το θέμα στη μερίσια διάταξη. Ε, Δυστυχώ η ίδια έπρεπε να πάει στην Ολλανδία και εγώ πρέπει να φύγω και εγώ πρέπει να πάω σε άλλη ε, επιτροπή. Γι' αυτό απλά εκ μέρου τη Έστερ Λάγκε ε, επιτρέψτε μου να σα διαβιβάσω ότι για την ίδια αυτό που προσθέτει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πώς ακριβώς σχετίζεται η οικονομική κρίση με τη φυματίωση, αν υπάρχει σχέση μεταξύ τους και τι ακριβώ γίνεται με την αντοχή στα ε, αντιβιωτικά, αντίδραστα αντιβιωτικά σε σχέση με τη θυματίωση. Ίσως μπορούν οι ομιλητές να τοποθετηθούν από αυτό. Ευχαριστούμε τον κύριο Λίζη ε, και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπερτολίνη. Παρακαλώ, κύριε Μπερτολίνη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είμαι εδώ εκ μέρου ε, του ε, ΠΟΗ. Θα ε, σα χαιρετίζει και ο Γενικός Γενικό Διευθυντή τη Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία. διαστόματός μου. Χαίρομαι όλους ιδιαίτερος που βρίσκομαι εδώ να συζητήσω μαζί σας το θέμα της πολυαμφιβητικής φυματίωσης στην Ευρώπη. Στις 26 Μαρτίου έχουμε την επέτειο της εφεύρεσης των την ανακάλυψη του βακίλου του Κόχ είναι ε, η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια πηγαίνει πέρα βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και πέρα από την ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο πηγαίνει και προς την πρώην Σοβιετική Ένωση, είναι πολύ ευρύτερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε 64 θανάτους στην περιφέρεια αυτή. Είναι ένας από τους μια μεγάλη αιτία θανάτου, ένα σοβαρός αριθμός ε, θανάτων. Ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ξενιστής ε, του μικροβίου και 10% του πληθυσμού, ε, αν ε, νοσή από την ασθένεια κατά τη διάρκεια της ε, ε, ζωής του. Πρόκειται λοιπόν για μια ασθένεια που μπορεί να θεραπευτεί, αλλά χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται δέσμευση και χρειάζεται και πολλή επένδυση από το σύστημα υγείας των διαφόρων χωρών. Δεν είναι ένα νέο πρόβλημα. Πλήττει την ανθρωπότητα εδώ και αιώνες υπήρχε και σε άλλες ε, υπήρους ε, και επειδή υπήρχε εμπόριο και μετανάστευση κυκλοφορούσε από τη μία ήπειρο στην άλλη. Δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό ότι η φυματίωση μειωνόταν ε, κατά τη διάρκεια της 19, του 19ου και του 20ου αιώνα πριν από την ύπαρξη αντιβιωτικών, πριν από την χρήση αντιβιωτικών στις θεραπείες και το συνδέω μάλιστα με το ερώτημα που ε, μόλις θέσατε για ε, τα, τις ε, συνθήκες διαβίωσης όπως επίσης και τις θρεπτικές συνήθειες. Για διάφορους λόγους η φυματίωση θεωρείται ένα ζήτημα του παρελθόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως δεν ισχύει, δεν είναι θέμα προηγούμενων γενεών. Είναι κάτι που επηρεάζει πολλά μέρη του κόσμου και την Ευρώπη και σήμερα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να λάβουμε ε, υπόψη ότι η φυματίωση δεν επηρεάζει τον καθένα και την κάθε χώρα με τον ίδιο τρόπο. Είναι κυρίως μια ασθένεια, off, ε, μια, ε, μια της φτώχειας. Επηρεάζει λοιπόν τους μετανάστες, τους φυλακισμένους. Να σας δώσω κάποια δεδομένα. 50% των γνωστοποιημένων κρουσμάτων στη Δυτική Ευρώπη είναι μεταξύ μεταναστών, ειδικότερα συγκεκριμένες χώρες και 2% των έγκλειστων ε, ε, σε φυλακές Ευρώπης ε, πάσχουν από φυματίωση. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να μην μας διαφεύγει. Ε, εν ώψη μάλιστα της ε, επιδείνωσης των οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων ε, σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτές οι οικονομικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν τις, τα συστήματα υγείας, την πρόσβαση στα φάρμακα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης φυματίωσης στα επόμενα έτη. Τώρα, το γεγονός ότι σήμερα, ακόμη και σήμερα, ακόμη και στη, στην τρέχουσα δεκαετία η φυματίωση είναι μεγάλο πρόβλημα, ε, δείχνει ότι ε, υπήρξε μεγάλο πρόβλημα ενδεχομένως και στη Δυτική Ευρώπη επειδή ε, στις αρχές της δεκαετίας του 90 κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, μειωνόταν στο τμήμα αυτό της Ευρώπης και σε άλλα μέρη της Ευρώπης η φυματίωση, όμως ξαφνικά άρχισε να αυξάνεται και πάλι. Και το γεγονός αυτό μαζί με άλλες τάσεις όπως για παράδειγμα ε, συνδυασμός φυματίωση και του ιού του AIDS και άλλου είδους αλληλεπιδράσεων ε, έγινε ένα, κατά κάποιο τρόπο φυσικό πείραμα ε, η επιδείνωση των οικονομικών και των κοινωνικών συνθήκων είναι ένας, ε, μια αιτία της φυματίωσης. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Σε 32 χώρες ε, ε, της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, περισσότερες των οποίων βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε σημαντική μείωση εμφάνισης νέων κρουσμάτων της ε, ε, ασθένειας σήμερα μιλάμε για ένα συνολικό πληθυσμό 210.000. Ε, ε, είναι σχετικά χαμηλός αριθμός. Γιατί υπάρχουν χώρες ε, που φέρουν το 85% του βάρους της φυματίωσης, κάτι το οποίο επηρεάζει την ευρωπαϊκή περιφέρεια γενικότερα. Στις χώρες αυτές 97% των ε, κρουσμάτων ε, έχουμε την ε, είναι η πολυανθεκτική φυματίωση. Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα είδος φυματίωσης το οποίο είναι ανθεκτικό σε δύο από τα πιο αποτελεσματικά αντιβιωτικά Refurbishing και Zonia Child ε, τα οποία βέβαια είναι πολύ ακριβά και όχι πάντοτε αποτελεσματικά. Αυτή λοιπόν η πολυανθεκτική φυματίωση ε, πλήττει ιδιαίτερα κάποιες χώρες της ε, περιφέρειάς μας και πάνω από το 30% των περιπτώσεων αφορούν περιπτώσεις που έχουν ήδη θεραπευθεί από φυματίωση στο παρελθόν. Εμφανίζεται και πάλι δηλαδή η ασθένεια το ίμιση των ε, ε, ασθενών αυτών μόνο μπορεί ε, που παρουσιάζουν την ασθένεια κατ' υποτροπή μπορούν και πάλι να θεραπευθούν με τη χρήση των αντιβιωτικών. Εξαπλώνονται με πολύ μεγάλους ρυθμούς η πολυανθεκτική φυματίωση. Επηρεάζει 15 από τις 27 χώρες και Μάλιστα, το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης νέων κρουσμάτων βρίσκεται ε, στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. 80.000 ε, κρούσματα, 80% δηλαδή του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων στην, ε, στον κόσμο. Γιατί? Γιατί ο αριθμός στην Ευρώπη είναι περίπου 5% του συνόλου. Δηλαδή μπορείτε να δείτε ότι για παράδειγμα, μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι τριπλάσιος ο αριθμός των κρουσμάτων από αυτό που θα περιμέναμε σε σχέση με το μέγεθος ε, της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Υπάρχει επίσης και μια περίπτωση ε, άκρος πολυανθεκτικής ε, φυματίωσης. 350 άτομα νόσησαν. Είναι ένα είδος φυματίωσης το οποίο είναι επίσης ανθεκτικό στο δεύτερο επίπεδο αντιβιωτικών. Επομένως είναι σχεδόν αδύνατη η θεραπεία. Ε, μπορεί ε, να θεραπευθεί σε μερικές περιπτώσεις, αλλά σε περισσότερες περιπτώσεις δεν θεραπεύεται. Είναι λοιπόν ε, ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο, γιατί χρειάζονται επιπλέον φάρμακα, επιπλέον θεραπεία, νοσοκομιακή περίθαλψη για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία. Ο ΠΟΗ ενώπιον αυτής της κατάστασης ε, κατά τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να ε, έχει ένα ενοποιημένο πρόγραμμα δράσης ε, το οποίο θα εφαρμόσει μέχρι το 2015. Έχει εγκριθεί από τους Υπουργούς Υγείας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκής Περιφέρειας τον περασμένο μήνα στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Μέχρι το 2015 θέλουμε να διαγνώσουμε τουλάχιστον το 85% των περιπτώσεων των κρουσμάτων πολυανθεκτικής ε, φυματίωσης. Δεν έχουμε βέβαια ακόμη τον πλήρη αριθμό. Μερικές φορές ε, ε, ο κόσμος πεθαίνει χωρίς να έχει πρόσβαση στη θεραπεία, ούτε καν στη διάγνωση. Οπότε 85% έχουν διαγνωστεί, 75% έχουν αποθεραπευθεί η εφαρμογή του σχεδίου δράσης, αν όντως γίνει στο πλαίσιο των χωρών, θα οδηγήσει σε πολύ ε, σημαντικά αποτελέσματα ε, θα οδηγήσει ε, σε 13.000, διάγνωση 13.000 τουλάχιστον κρουσμάτων άκρος πολυανθεκτικής, πολυανθεκτικής φυματίωσης και περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής θα εξοικονομηθούν. Ε, χρειάζεται μια επένδυση 5 δισεκατομμυρίων, αλλά αν αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι τεράστιο το κόστος, επομένως έχει κάποιο νόημα ε, αν δει κανείς την ανάλυση του κόστους και του ωφέλους ε, να γίνει επένδυση αυτή. Θα σώσουμε και χιλιάδες ζωές. Είναι λοιπόν δύσκολο βέβαια κανείς να ποσοτικοποιήσει την αξία της ζωής, την τιμή της ζωής, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, εμένα μου είναι κάθε φορά πολύ δύσκολο να κάνω τέτοιου είδους αναλογίες. Είναι κάτι όμως το οποίο πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. ο ΠΟΗ έχει δεσμευθεί να ε, βοηθήσει και ε, τεχνικά τις χώρες ώστε να εφαρμόσουν το ε, πρόγραμμα αυτό και αυτό μπορεί να γίνει σε πολλές πτυχές. Υπάρχει η πτυχή της έρευνας γιατί χρειαζόμαστε για την άκρος πολυανθεκτική φυματίωση νέα φάρμακα αλλά υπάρχει και η πτυχή της θεραπείας και της πρόληψης. Και όταν λέω πρόληψη εννοώ και τον επαρχή έλεγχο, έλεγχο της εξάπλωσης της ασθένειας. Γιατί υπήρξαν πολλές περιπτώσεις σε κάποιες χώρες τη ε, Ευρώπη ότι ε, σε... Ε, ε νηπιαγωγία που εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα η ασθένεια. Και πρέπει να δούμε επίση και τι χρηματοδότηση υπάρχει. Υπάρχει ένα παγκόσμιο ταμείο για τη φυματίωση, την ελονοσία και το AIDS που ε, δεν θα χρηματοδοτήσει ε, μέχρι το 2014. Υπάρχει λοιπόν τεράστια έλλειψη πόρων και γι' αυτό πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ε, αντιμετωπίσουν αυτό το, το, αυτό το ζήτημα. Γιατί η ανεπάρκεια ε, των πόρων μπορεί να οδηγήσει σε ε, ακόμη μεγαλύτερη εξάπλωση της ασθένειας σε ε, βαθμό που μπορεί να υπάρξει πλήρης ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά και θα έχουμε ένα πρόβλημα του πώς να αποθεραπεύσουμε τους ασθενείς. Συνοψίζω λοιπόν τώρα. Ποια είναι τα μηνύματα που θα ήθελα να λάβετε σήμερα η φυματίωση δεν είναι μόνο θέμα αναπτυσσόμενων χωρών ή κάποιων τμήματων της Ευρώπης, αλλά όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, είτε άμεσα είτε έμεσα λόγω μετανάστευσης από άλλα μέρη του κόσμου, λόγω ορισμένων τμήματων του πληθυσμού που είναι πιο ευπαθή λόγω της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Δεύτερο μήνυμα. Η πολυανθεκτική φυματίωση είναι μεγάλος ε, κίνδυνος μεγάλη απειλή, μπορεί να θέσει ένα κινδύνο την πρόοδο που σημειώθηκε του τελευταίου αιώνε, καθώ και τη δυνατότητα μελλοντική θεραπεία. Τρίτον, η οικονομική κρίση αυξάνει τον κίνδυνο. Είναι ένα πλαίσιο που μπορεί να αντιστρέψει τη σημειωθήσα πρόοδο και να μειώσει τη δυνατότητα ελέγχου της ασθένεια Και τελευταίον, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις για τον έλεγχο και τη θεραπεία και στην Ευρώπη και στις γειτονικέ περιοχές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπερτολίνη για την ομιλία σας. Και τώρα η Επιτροπή, την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Τζον Ράιν, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δημοσίας Υγείας, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Όσο προσεγγίζουμε την Παγκόσμια ημέρα για τη φυματίωση, ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας για την οργάνωση αυτής της συνάντησης. Όπως ακούσαμε από τους συναδέλφους του ΠΟΗ, η φυματίωση εξακολουθεί να είναι σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε όλη την Ευρώπη αλλά και σφαιρικά. Γνωστοί οι λόγοι. Χαμηλό ποσοστό θεραπείας έχει εξαπλωθεί η ανθεκτική στα φάρμακα οι μειονεκτικές ε, πτυχές της κοινωνίας δεν έχουν δυνατότητα να αντιμετωπίσουν και έχουμε βεβαίως και τη μεγάλη πρόκληση σε πολλά κράτη-μέλη που δημιουργεί η οικονομική κρίση. Έναντι αυτή τη κατάσταση, η Επιτροπή έχει αναπτύξει μια πολιτική και οικονομικές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε τη φυματίωση και την πολυθεκτική φυματίωση όσον αφορά την έρευνα, την επιτήρηση, την πρόληψη και τον έλεγχο και η διεθνή συνεργασία. Στον τομέα της έρευνας, η, Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει το τρίτο πρόγραμμα πλαισίου, νέες μεθόδους διάγνωσης, πάνω από 125 εκατομμύρια ευρώ έχουμε δαπανίσει για την έρευνα για τη θυματίωση τα τελευταία 10 χρόνια. Υποστηρίζουμε, για παράδειγμα, την πρωτοβουλία για εμβολιασμό κατά τη θυματίωση που, που λειτουργεί από το 2008 ως εταιρική σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οι ευρωπαϊκές και οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μια εταιρική σχέση για κλινικές δοκιμές που χρηματοδοτήθηκαν από 60 εκατομμύρια για κλινικές δοκιμές από το 2008 για βελτιωμένα ή νέα φάρμακα, διαγνωστικές μεθόδους και εμβόλια στην υποσαχάρια Αφρική με βάση το σχέδιο δράσης του προγράμματος πλαίσιο κατά της φυματίωσης χρηματοδοτούμε προγράμματα για να αυξήσουμε τη δυνατότητα των κρατών μελών πρόληψης και καταπολέμησης της φυματίωσης. Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα για τη βελτίωση του ελέγχου για τη διάγνωση σε περιθωριοποιημένα τμήματα της κοινωνίας, την ενίσχυση της επιτήρησης για τη φυματίωση στην Ευρώπη και την αύξηση της ορατότητας και της συνειδητότητας του κινδύνου φυματίωσης στον πληθυσμό. αυτέ οι προσπάθειέ μας για την πρόληψη και έλεγχο της φυματίωσης θα ενισχυθούν περαιτέρω από μια πρόσφατη κοινοτική πρωτοβουλία πέρυσι το Νοέμβριο για να αντιμετωπίσουμε την ε, πολυανθεκτική φυματίωση. Το σχέδιο δράσης 11-15 για την αντιμετώπιση της αντίστασης στα μικρόβια θα ασχοληθεί και με αυτή την ασθένεια για να αναπτύξουμε νέα, πιο αποτελεσματικά αντιβιωτικά, νέε μεθόδου θεραπεία και καλύτερε μεθόδου διάγνωση Οι προσπάθειε. Αυτέ δεν περιορίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζουμε και τι αναπτυσσόμενες χώρε στι προσπάθειε του να βελτιώσουν την υγεία των κατοίκων του και να αντιμετωπίσουν μεγάλε σοβαρέ ασθένειε, όπω η φυματίωση. Ήδη από το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δαπανίσει περίπου ένα δις για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. Υπάρχει όμως και σε κάποια κράτη της Ένωσης, όπως Βουλγαρία και Ρουμανία. Εδώ χορηγούμε πάνω από 60% της ε, διεθνούς βοήθειας για αντιμετώπιση. Αυτές οι προσπάθειες για διεθνή συνεργασία, πρόληψη και έλεγχο αποδεικνύουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σφαιρική αντιμετώπιση της φυματίωσης. Μαζί με αυτές τις ενέργειες να δούμε και τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που ευνοούν την νόσο. Πρέπει επίση να κινητοποιήσουμε όλα τα όργανα που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα αίτια. Η υγεία, για παράδειγμα, είναι σημαντικό προσόν για την περιφερειακή ανάπτυξη. Εάν επενδύσουμε στη φροντίδα για τους ασθενείς, την περίθαλψη και την πρόσβαση στην υγεία για τις ε, ευπαθείς ομάδες, την πρόληψη των ασθενειών, την εκπαίδευση, και την κατάρτιση των επαγγελματιών τη υγεία βοηθάμε την περιφερειακή ανάπτυξη και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό και Ταμείο Συνοχή από το 2007. Δεν αντιμετωπίζουμε έτσι απευθεία την εφηματίωση, αλλά ενισχύουμε τα εθνικά συστήματα υγεία, τη δυνατότητα καταπολέμηση των ε, μεταδεδομένων των ε, ασθενειών, όπω η εφηματίωση. Το Ταμείο Συνοχή λοιπόν μα βοηθά να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση της καταπολέμησης της ασθένειας στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Βεβαίως πρέπει να τροποποιηθούν και να μεταρρυθμιστούν τα συστήματα υγείας. Έχουμε επίσης ε, και υπάρχει επίσης ανάγκη να υπάρξουν και πολυτομεακές προσεγγίσεις. Πρέπει να εργαστούμε στενά με όλους τους εμπλεκόμενους. Τα τελευταία χρόνια στόχος μας ήταν να βελτιωθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις προσπάθειες κατά της φυματίωσης και σε συνεργασία με το ECDC και τον ΠΟΗ δώσαμε μια σειρά από βραβεία σε μη κυβερνητικές οργανώσεις για να αυξηθεί η ορατότητα της συμμετοχής τους. Το 2010 οργανώσαμε μαζί με το ECDC μια δημόσια διαβούλευση στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου καταπολέμησης και το 2011 το πρόγραμμά μας για την υγεία προέβλεπε μια νέα πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της ε, φυματίωσης με την εμπλοκή και των δημοσίων αρχών και της κοινωνίας των πολιτών για να εμπλέξουμε τις ευπαθείς ομάδες. Η φυματίωση είναι τομέα κλειδί στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον ΠΟΗ. Με βάση αυτή την ήδη υπάρχουσα συνεργασία, ελπίζουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας. Γιατί αυτή η νόσο σίγουρα δεν σέβεται σύνορα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα λοιπόν ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στον διδί του ECDC, τον κύριο Σπραγκιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε εδώ. Ε, θα ήθελα κανονικά να σας δώσω και ευχάριστες και αρνητικές ειδήσει, έτσι να υπάρχει μια ισορροπία, αλλά είναι δύσκολο να σας αναφέρω και ευχάριστες ειδήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ECDC. Είχαμε ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουμε την πολυανθεκτική θυματίωση. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο τελικά. Αν έξω μια ματιά στα τελευταία πέντε χρόνια, το μόνο που επιτύχαμε ήταν μια μικρή μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων πολυανθεκτικής θυματίωσης. Ε, Και αυτά τα καλά χρόνια. Τότε δηλαδή που ε, διατέθηκαν ε, αρκετά κονδύλια. Όμω, δεν είμαι αισιόδοξο για τα επόμενα χρόνια γιατί θα έχουμε λιτότητα, δεν θα υπάρχουν πια οι παχέ και γιατί είμαι απεσιόδοξο διότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στην Ευρώπη σημαίνει κατ' ουσίαν δύο πράγματα. Πρώτον, περικόπτονται οι προπολογισμοί υγεία και δεύτερον και περισσότερο όλο και περισσότεροι άνθρωποι εξωθούνται στην ε, εξατλίωση. Αυτοί λοιπόν ε, δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν ε, τη θυματίωση, όπως αναφέρθηκε και από τον ΠΟΕ. Η φτώχεια είναι η ασθένεια των φτωχών, σπάνια η μεσαία τάξη προσβάλλεται από όσο για τους πλούσιους αυτοί δεν προσβάλλονται ποτέ. Όμω, η φυματίωση εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρυσι περίπου 74.000 κρούσματα καταγράφηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων περίπου 1.500, 1500 περιπτώσεις ήταν πολυανθεκτικά κρούσματα. Συνήθω είπαμε οι φτωχοί, οι περιφερειοποιημένοι, οι μετανάστες, ε, οι έγκλησες φυλακέ, οι Ρώμα, ε, οι άστεγοι, οι φτωχοί γενικότερα στις πόλεις. Αυτές λοιπόν οι ομάδες, οι περισσότερο ευπαθείς ομάδες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθώς ε, συνεχίζεται η οικονομική κρίση, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι θα διολυστήσουν σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Όλο περισσότερο άστεγοι, περισσότερο έγκλημα, εθισμοί, αλκοολικοί. Δεν είναι αισιόδοξη λοιπόν η εικόνα. Και γι' αυτό θα αυξάνεται ο ευπαθής πληθυσμός. Πάντως ε, θα πρέπει να εκταμιευτούν πόροι για να αντιμετωπιστεί η φυματίωση. Δύσκολο αυτό. Όλο και πιο δύσκολο. Και χρειαζόμαστε όλο και περισσότερους πόρους. Γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά. Γιατί είναι δύσκολο να διαγνωστεί η φυματίωση και δύσκολο και να αποθεραπευτεί. Άρα δηλαδή μιλάμε για μια περίπτωση που χρήζει πολλών πόρων. Ξέρετε ποια είναι τα κλασικά συμπτάντα της ε, ευματίωσης, κούραση, ε, βήχας, ε, κόπωση. Αυτό αυτά τα συμπτώματα προσφέρονται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και ο γιατρός ο μόνος τρόπος για να είναι σίγουρος ότι ο ασθενής πάσχει από πρέπει να προβεί σε εργαστηριακές δοκιμές με τα σωστά μηχανήματα να υπάρχει και σωστή γνώση διάγνωσης άρα και μόνο η διάγνωση είναι δαπανηρή Ποια είναι λοιπόν και τα συμπτώματα της ε, πολυαντεκτικής ε, Φα... Δεν διαφέρουν από την κανονική θυματίωση. Ο μόνος τρόπος για να τη διαγνώσει κανείς είναι να γίνουν συμπληρωματικές ε, διαγνωστικές μελέτες. Η διάγνωση αυτής της πολυαντεκτικής θυματίωσης απαιτεί και περισσότερες γνώσεις και πολύ καλά εξοπλισμένα εργαστήρια. Έχουμε λοιπόν στο δικό μας ε, το κέντρο πολλά εργαστήρια που στηρίζουμε. Έχουμε καταβάλει πολλές προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η πολυανθεκτική ε, φυματίωση και έχουμε διαδώσει γνώση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα εργαστήρια. Όμως ε, τα εθνικά τα εθνικά κέντρα στηρίζονται από τα κράτη-μέλη και εάν περικοπούν οι επιδοτήσεις για τα εργαστήρια και για το προσωπικό δεν θα μπορούμε να προβούμε σε διάγνωση της απλής μα πόσο μάλλον της πολυαντεκτικής. Άρα θα υπάρχει καθυστερημένη διάγνωση και τι σημαίνει αυτό ότι ε, θα διαδίδεται όλο και περισσότερο ευματίωση. Ξέρετε πόσο καιρός χρειάζεται για να ε, θεραπευτεί ένα κρούσμα. Έξι μήνες αν έχει κανείς την απλή θυματίωση, αλλά δύο χρόνια αν έχει κανείς προβληθεί από την πολυαντεκτική. Ε, το ε, πρωτόκολλο της θεραπείας είναι περίπλοκο, ε, χρησιμοποιούνται τέσσερα διαφορετικά αντιβιωτικά τους δύο πρώτους μήνες και δύο διαφορετικά αντιβιωτικά για τους αναπομένοντες τέσσερις μήνες. Όλα αυτά είναι δαπανηρά. Η θεραπεία για την πολυαντεκτική θυματίωση χρειάζεται και ενσυνδεμένη με περισσότερα φάρμακα. Πάντως η θυματίωση και η πολυαντεκτική πρέπει να είναι υπό την παρακολούθηση επαγγελματιών, γιατί αλλιώς αν η απλή δεν διαγνωστεί σωστά, θα γίνει πολύ ανθεκτική. Κατόπιν τούτου, γι' αυτό εμφανίζεται αυτή η φυματίωση. Η απλή φυματίωση χρειάζεται λοιπόν πόρους για τα εργαστήρια, για φάρμακα, ε, τους για να ελέγχουν τη θεραπεία και χρειάζεται βέβαια και εθνικά Ινστιτούτα για να ελέγχουν και να αξιολογούν ε, τη θεραπεία. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι αν όλα γίνουν κατά γράμμα και αν καταλήξουμε σε πολυανθεκτική θυματίωση μόνο το 30% των κρουσμάτων θα αποθεραπευτεί. Που δεν είναι σωστό, δεν είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Πρέπει να σας πω, εγώ δεν είμαι πεπισμένο ότι όλα τα κράτη-μέλη θα εκταμιεύσουν τους απαραίτητους πόρους για να ελέγχεται η θυματίωση κατά τα επόμενα έτη. Ε, και αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο μάλλον για τις χώρες της Ασίας, ε, όπου οι όροι που ε, εκταμείονται είναι ακόμα λιγότεροι. Οι ευρωβουλευτέ αλλά και οι εθνικοί βουλευτέ μπορούν όμω να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο έτσι ώστε ο έλεγχο συμματίωση ε, να έχει την προτεραιότητα που του αξίζει. Η ΟΠΟΕ και το δικό μα το Ευρωπαϊκό Κέντρο θα συμβάλλουν, ε, θα στηρίξουμε και εμεί τι δεσμεύσει σα. Ας δούμε λιγάκι πόσα κρούσματα παρουσιάστηκαν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρυσι. Αν δει κανείς ε, την εμφάνιση αυτών των νέων κρουσμάτων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολλέ και μεγάλες διαφορέ. Η εμφάνιση ε, νέων κρουσμάτων είναι ανά χίλιους κατοίκους. Και έτσι μπορεί κανείς λιγάκι να συνέχει συμπεράσματα για το κατά πόσο υπάρχει επιδημία φυματίωση σε μια χώρα. Βλέπουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε λιγότερα νέα κρούσματα απλή φυματίωσης και πολυανθεκτικής από ό,τι σε άλλες περιοχές. Σε 21 κράτη-μέλη θεωρούμε ότι είναι χώρες με λίγα νέα κρούσματα, δηλαδή ε, λιγότερες ε, από 20, από 20 κρούσματα σε χίλιους. Και έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μείωση. Όμως, αν δούμε λιγάκι την τάση ε, της πολυανθεκτικής θυματίωσης τα τελευταία πέντε χρόνια, καταλήγουμε στο ότι η τάση είναι επίπεδη. Αν όμως το δει κανείς πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι η ακραία θυματίωση θα αυξηθεί κατά τα επόμενα έτη. Και η χώρα, η εικόνα στις χώρες με χαλμηλή εμφάνιση νέων κρουσμάτων δεν είναι τόσο καλή. Γιατί ε, υπάρχουν κάποιοι υψηλής ε, Εμφάνιση. Έχουμε λοιπόν κάποια καλά νέα, αλλά όπως σας είπα έχουμε και θύλακες φυματίωσης στις μεγάλες πόλεις. Μία ε, μελέτη που έγινε κατέδειξε Λονδίνο, Παρίσι, Κοπεχάγη, Ρότερνταμ, τέτοιου είδους πόλεις έχουν τριπλάσια εμφάνιση κρουσμάτων θυματίωση και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, να εξαλειφθεί η θυματίωση σε αυτές τις πόλεις. Πενταπλάσια τα κρούσματα στην, στο Μιλάνο σε σχέση με την υπόλοιπη Ιταλία και ο λόγος η φτώχεια. Ή στις μεγάλες πόλεις έχουμε συνήθως περισσότερους άστεγους, ε, νέου ε, νέους μετανάστες και Ξέρουμε, α πούμε, την περίπτωση τη Νέα Υόρκη. Έχει περάσει βέβαια κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά η Νέα Υόρκη απέδειξε ότι αν δεν αποδώσουμε σημασία στον έλεγχο τη ματίωση, κάποια στιγμή αργότερα θα ξεσπάσει η ασθένεια αυτή. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι οι πόροι για την φυματίωση μειώνονται και αυτό μοιάζει να είναι αισιόδοξο. Βεβαίω, αν δεν έχει κανεί κρίματα για να κάνει τη διάγνωση, προφανώ και δεν εντοπίζει νέα κρούσματα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Θέλει προσοχή. Σημαντικό είναι να υπάρχει καταρχήν διάγνωση και μετά η θεραπεία. Αν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια, διαπιστώνουμε ότι τελικά θα εμφανιστεί έξαρση της ασθένειας μετά από κάποια χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν τελειώνοντας θέλω να σας καλέσω αύριο στο Λονδίνο και την Παρασκευή στη Βαρκελόνη, το Ρότερνταμ και το Μιλάνο. Εκεί θα έχουμε εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα της ευματίωσης. Εγώ θα πάω στο Ρότερνταμ και σε κάθε μία από αυτές τις εκδηλώσεις θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην αστική φηματίωση οι πόλει που διοργανώνουν αυτές τις εκδηλώσεις θα χαιρόντουσαν πάρα πολύ αν μπορούσατε να τι βοηθήσετε και να τις στηρίξετε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σπρέγκα για την παρουσίασή σας και κατανοήσαμε πόσο δραματική είναι η εικόνα. Πρέπει πράγματι να κινητοποιηθούμε για αυτό το θέμα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο ε, στους αδέλφους, πρώτη κυρία Ροσπάχ. Άννα Ροσπάχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω, να καλωσορίσω τους εκπροσώπους ε, από τον ΠΟΗ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το ECDC και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συζητήσουμε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Για μένα μια τόσο τρομακτική ασθένεια όπως η φυματίωση το να ε, παρουσιάζεται και να αυξάνεται η εξάπλωσή της ε, είναι τρομερό. Είναι πραγματικά ένας ε, κίνδυνος για την υγεία των πολιτών στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω ορισμένα ερωτήματα είδα την ε, παρουσίασή σας ε, και έχετε κάποια στοιχεία σε σχέση με, τα, με το κόστος ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, θεωρεί, πόσο, πόσο νομίζετε ότι κοστίζει η πολυανθεκτική φυματίωση στην Ευρώπη. Έχετε στοιχεία και επίσης το να μην κάνουμε τίποτε τι θα μας κοστίσει. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Θα ήθελα επίσης ε, να μάθω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τι έχουμε ήδη κάνουμε για να προλάβουμε την εξάπλωση και τη απλή, αλλά και της πολυανθεκτική φυματίωση. Και θα ήθελα να, να δω αν έχουν ληφθεί συγκεκριμένα ε, βήματα στις χώρες για το θέμα αυτό. Οι αρχές, ε, ε, οι αρχές στα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει δεσμεύσεις επί του ζητήματος αυτού και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν ε, ε συλλέγετε τις βέλτιστες πρακτικές από τις, άλλες, από τις διάφορες χώρες ή από άλλους οργανισμούς στο ECDC, όπως κάνει ο ΠΟΗ, για παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Λίντα Μακάβαν. Um, Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που το συζητούμε σήμερα. Είχα πάει στην Ουκρανία πριν από μερικά χρόνια με μια μη κυβερνητική οργάνωση που λεγόταν Results και συζητούσε, εξέταζε τη φυματίωση σε αυτό το τμήμα ε, της ε, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σε φυλακές της Ουκρανίας και σε νοσοκομεία τότε οι γιατροί που είχαμε συναντήσει μας είχαν πει ότι η κατάρρευση του συστήματος υγείας ε, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ε, ο βασικός λόγος γιατί δεν υπήρχε πρόσβαση πλέον τόσο μεγάλη σε φάρμακα. Ξέρουμε ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκαν ε, η μείωση, ε, οι περικοπές ε, στο σύστημα υγείας. Στην Ελλάδα, βλέπουμε τι προβλήματα υπάρχουν ε, με τις περικοπές στο σύστημα υγείας και στην Πορτογαλία υπάρχουν προβλήματα με τις πληρωμές των γιατρών. Ξέρω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και στη Ρουμανία για την πρόσβαση στα φάρμακα. Είναι ζητήματα λοιπόν που θα έπρεπε να μας απασχολούν και να το σκεφτούμε ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τα προγράμματα λιτότητας. Μπορούμε να γνωρίζουμε τώρα τι θα πει, που μπορεί να καταλήξει η λιτότητα και πρέπει να το έχουμε κατά νου ε, όταν ε, μιλάμε για περικοπές ε, ακόμη και στα συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Θα ήθελα να θέσω λοιπόν τα σχετικά ερωτήματα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο ECDC. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη πώς συνεργάζεστε. Δεν κατάλαβα ποιος δρομολόγησε αυτό το σχέδιο δράσης πέρσι. Αναφερθήκατε σε κάποιο πριν από μία πενταετία, αλλά αναφέρατε και ένα καινούριο και θα ήθελα να μάθω αυτό το σχέδιο δράσης πώς λειτουργεί και τι ακριβώς ε, επιζητά από τα κράτη-μέλη. Θέλουν χρήματα γιατί ε, υπόθηκαν κάποια πράγματα για τα ερευνητικά προγράμματα και για τα σχέδια δράσης για την υγεία, αλλά δεν έχω καταλάβει πολύ καλά το νέο πρόγραμμα, εάν απλώς ε, ε είναι ένα επιστέγασμα όλων των υπολείπων ή αν είναι κάτι ακόμη. Ε, είπαμε ότι θα ξοδέψουμε δισεκατομμύρια ευρώ αν δεν κάνουμε τίποτε γι' αυτό, αλλά πείτε μας πόσα χρήματα χρειαζόμαστε. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμμετέχει σε μια προσπάθεια ε, εξέβρεσης χρηματοδότησης. Τι θα κάνουμε ακριβώς, απλώς ο κόσμος θα υποβάλει σχέδια δράσης και μετά θα ελπίζουμε ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση. Υπάρχει λοιπόν κάποιο κάποια συνοχή, κάποια συνοχή σε όλες αυτές τις προσπάθειες, με όλα αυτά τα προγράμματα και τα κονδύλια που χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σίγουρα μεγάλη πρόκληση, λέει η κυρία Σάλτεμος. Χρειάζεται περισσότερη δράση στον τομέα αυτό. Βεβαίως είναι δύσκολο να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Γι' αυτό απευθυνόμενοι στην Επιτροπή. Αναφέρατε πολλές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναλυφθεί, έρευνα και άλλες πρωτοβουλίες. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε πρόβλεψη με βάση τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει. Πότε θα υπάρξει ουσιώδης μείωση των νέων κρουσμάτων απλής και πολυανθεκτικής φυματίωσης. Και προς τον Δόκτωρα Σπρίγκερ και τον Πόη θα ήθελα να μάθω. σε πόσο καιρό πιστεύετε ότι θα επανέλθουν, θα επανακάμψουν οι επενδύσεις στον τομέα αυτό σε 2, 3 ή σε 10 χρόνια. Γιατί αυτό πρέπει να μας αφορά και εμάς ως πολιτικούς. Ανησυχητικά νέα αυτά που μας φέρατε, αλλά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κρίστολ. Τανέσκου παρακαλώ. Και Κεντά Μέρκης. Όπως αποδεικνύει το πρόγραμμα δράσης του ΠΟΗ, πρέπει να αντιμετωπίσουμε επιγόντως και στην Ευρώπη την πόλη ανθεκτική φυματίωση. Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις για τις τρεις ασθένειες που προαναφέρθηκε δίνουν χρηματοδότηση επαρκή αυτή τη στιγμή για την καταπολέμηση της ασθένειας αυτήν στην Ρουμανία. Αλλά είπατε ότι για την επόμενη περίοδο δεν θα υπάρχουν επαρκή χρήματα μέχρι το 2014. Οπότε θα υπάρξουν σοβαρές περικοπές και δεν θα είμαστε σε θέση να καταπολεμήσουμε την ε, πολύ φυματίωση. Οπότε, ρωτάω, Πώς θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις χώρες που θα έχουν τέτοιο κενό χρηματοδότησης και τι προοπτικές υπάρχουν να επανέλθει αυτή η χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Μέρκης παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τα πολύ ενδιαφέροντα και ανησυχητικά βέβαια αυτά που μας ε, είπαν. Σοκαρίστηκα ακούγοντας ότι στη δική μου τη χώρα εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα όχι μόνο υφέρπει, αλλά έχει ξεσπάσει. Επειδή λοιπόν πρόκειται για μια ασθένεια που έχει σχέση με τη φτώχεια και επειδή βλέπουμε ότι η φαρμακευτική βιομηχανία δεν επενδύει τόσο σε ε, φάρμακα που έχουν σχέση με τη φτώχεια, α το πούμε έτσι απλά. Εσείς μπορείτε να τους πείσετε να επενδύσουν σε ένα τομέα που ενδεχομένως δεν θα έχουν το ίδιο κέρδο. Να το πω με άλλα λόγια. Ε, διαπιστώσαμε ότι μόνο 15 εταιρείε ε, αυτή τη στιγμή επενδύουν σε ε, μικροβιωτικά Πώς μπορούμε λοιπόν να δώσουμε κίνητρα στη φαρμακευτική βιομηχανία για να ε, επενδύσει σε φάρμακα για την πολυαντεκτική χρηματίωση. Και όσον αφορά τα αντιβιωτικά, ε, είναι πολύ δύσκολο να γίνει και σύγκριση των στοιχείων, γιατί σε μία χώρα υπάρχει υπερβολική χρήση, κατάχρηση αντιβιωτικών, ενώ σε άλλες χώρες πάλι ε, μεγάλη επιφύλαξη. Πολύ διστακτικά ε, συνταγογραφούνται τα αντιβιωτικά. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, μπορούμε να κάνουμε τελικά μια πραγματική σύγκριση στην Ευρώπη για τα φάρμακα και για τις συνήθειες χορήγησης και χρήσης ε, φαρμάκων. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Άλλος παρακαλώ. Ποιος θέλει ε, πρώτος να απαντήσει. Παρακαλώ. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένες από τις ερωτήσεις που ετέθησαν και με τη σειρά που υποβλήθηκαν. Πρώτον, όσον αφορά ε, το κόστος της πολυαντεκτικής θυματίωσης. Έχουμε υπολογίσει ότι περίπου 50.000 ευρώ σε δύο χρόνια για άτομα που πρέπει να διακομιστούν σε νοσοκομείο για τρεις μήνες. Αυτό δεν ε, είναι σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια. Μερικοί πρέπει να ε, ενταχθούν στο νοσοκομείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάλογα με το πώς αντιδρούν στην ασθένεια. Και στις περιπτώσεις αυτές το κόστος ανεβαίνει στα 100.000 ευρώ ανάτομο. Είναι λοιπόν σημαντικό το κόστος. Και όπως είπα και στην ομιλία μου, έχουμε υπολογίσει ότι σε γενικές γραμμές ε, έχουμε επένδυση 5 δις ε, για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης. Αυτό θα απέδιδε 7 δις σε σχέση με το κόστος 12 δις που θα ήταν το κόστος της αδράνειας, του να μην κάνουμε τίποτα δηλαδή. Και όλες τις άλλες ε, συνέπειες τα συνεπακόλουθα. Όσον αφορά τώρα στη συνεργασία με το κέντρο η e ε, Σίγουρα ο συνάδελφος θα πει περισσότερα, αλλά να σας πω ε, και εγώ κάτι. Πρόκειται για ένα σύστημα ελέγχου που εφαρμόζουμε από κοινού με το κέντρο αυτό και ένας αποτελεσματικός τρόπος για να χρησιμοποιούμε τους πόρους. Αποφεύγουμε επικαλύψεις, ε, προχωράμε συντονισμένα. Όσον αφορά τώρα στο ερώτημα στη σχέση ανάμεσα στην οικονομική κρίση και την αύξηση των κρουσμάτων στις πρώην χώρες Σοβιετικής Ένωσης μετά το 1990, υπάρχει αυτό το γράφημα που δείχνει με απόλυτη σαφήνεια την αύξηση του αριθμού κρουσμάτων στην οποία στην περίοδο κατά την οποία υπήρχε αναταραχή και έτσι υπήρχε και ευνοϊκό περιβάλλον για την έξαρση της ασθένειας. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα μέτρα, γιατί μερικές φορές ε, πρέπει να πω ότι δυστυχώς τα μέτρα ε, είναι βραχυπρόθεσμα. Ξεχνάνε δηλαδή ποιες είναι μακροπρόθεσμες ε, συνέπειες και το κόστος. Γιατί μερικές φορές τους υπολογισμούς που γίνονται δεν λαμβάνεται υπόψη το μακροπρόθεσμο κόστος ορισμένων μέτρων. Όσον αφορά τώρα στο πρόγραμμα δράσης, ε, περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που ξεκινούν από τη βελτίωση της διάγνωσης με μοριακές διαγνωστικές τεχνικές. Υπάρχουν και κάποιες άλλες τεχνικές οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον ΠΟΕ και επιτρέπουν τον εντοπισμό κρουσμάτων με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι κατά το παρελθόν. Ε, κοστίζουν περίπου 40 ευρώ ε, το τεστ, αλλά αξίζει τον κόπο, διότι επιταχύνει τον εντοπισμό κρουσμάτων. Ε, από ημέρες ε, πάμε σε διάγνωση μέσα σε ορισμένες ώρες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η βελτίωση. Πάντως, αν θέλετε, μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες και μπορώ και εγώ να σας αναφέρω το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου φαίνονται με απόλυτη ακρίβεια οι διάφορες δράσεις μας. Συνεργαζόμαστε με το κέντρο και τις χώρε για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα. Όλα αυτά βέβαια απαιτούν χρηματοδότηση και όπως πολύ σωστά επισημάνατε ορισμένοι από εσάς, ε, υπάρχει πρόβλημα ε, οικονομικό σε ορισμένε χώρε. Ε, το ανέφερε ο συνάδελφο από τη Ρουμανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα. Και μερικέ φορέ αποκτά κανείς κάποια σημαντικά αποτελέσματα και έχει το αίσθημα ότι κάτι γίνεται. Άλλες φορές πάλι δεν υπάρχουν χρήματα και δημιουργείται υποτροπιασμός, προκαλείται υποτροπιασμός. Τώρα, όσον αφορά το πότε θα ξαναγίνουν επενδύσεις, κοιτάξτε, δεν απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας για την περίοδο 11 έως 15 και η εφαρμογή του προγράμματος δράση σε όλες του τις πτυχές θα μπορούσε να αποδώσει 250.000 κρουσμάτων ε, που θα διαγνωστούν. Σημαντικό αυτό, όπως είπε και ο Μάρκος, ε, γιατί είπε και εκείνο υπάρχει υπηματίωση όσο, ε, όσο γίνεται διάγνωση, αλλιώς μπορεί να πει και δεν υφίσταται. 120 τόσες χιλιάδες ζωές σώθηκαν Άρα δηλαδή αυτό είναι μια σημαντική απόδοση και μπορεί να μετρηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ποσοτικά και θα πρέπει βέβαια όλο αυτό να αποδοθεί στο πρόγραμμα δράση, στο βαθμό που εφαρμόζεται. Γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά, όπου δεν υπάρχει καμία παρέμβαση και εκεί τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα αρνητικά. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο, τον δόκτωρα Μπερτολίνη και θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στις ερωτήσεις ε, που Ετέθησες. Κύριε Ράιν, να ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Ε, για το πρώτο θέμα, κατά πόσο δηλαδή τα κράτη-μέλη παίρνουν σοβαρά την αφηματίωση. Είναι υποχρεωμένα να την πάρουν σοβαρά, γιατί είναι μία από τις μεταδιδόμενες ασθένειες που καλύπτεται από την νομοθεσία μας. Από το 1988 ε, ε, έχουμε νομοθεσία για τις μεταδιδόμενες ασθένειες και αναφέρεται μεταξύ αυτών και η φυματίωση. Δεν είναι η μόνη που καλύπτεται, γιατί ακούσαμε ότι υπάρχει και το θέμα της, αντί, της αντοχής στα, στα αντιβιωτικά ε, ότι είχαμε αυτή την εβδομάδα μία συνεδρίαση των κρατών μελών για να αποφασίσουμε για ε, τους ορισμούς της ε, ε, ε μικροβιακής ε, αντοχής και ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να μας ενημερώνουν όταν υπάρχουν ε, επιδημίες φυματίωσης ή άλλων είδο, άλλου είδους αντίστασης ε, σε ε, αντιβιωτικά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερον, η νομοθεσία αυτή υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να συλλέγουν και να υποβάλουν ετησίως στο ECDC στατιστικές. Επομένως, έχουμε συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε σύν χρόνο. Δεύτερον, όσο το, όσον αφορά το θέμα του Παγκοσμίου Ταμείου, πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολούθησε ε, την ε, αναθεώρηση του πάνελ υψηλού επίπεδου, ε, επιβεβαιώνοντας ότι είχαν υπάρξει κατάλληλα μέτρα για την μείωση σε σημαντικό βαθμό του κινδύνου στο μέλλον, όπως επίσης και την περίπτωση εντοπισμού απατών. Και βάσει των συστάσεων λοιπόν του Παγκοσμίου Ταμείου, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να ε, δώσει 330 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2011 έως 2013. Επομένως, ε, είχαμε ε, συζητήσει το, τα προβλήματα που υπήρχαν με το σύστημα ε, ελέγχου από κοινού με το Παγκόσμιο Ταμείο και καταλήξαμε σε, ε, στην υπόσχεση για αυτό το ποσό. Όσον αφορά τώρα την πολιτική συνοχή για την υγεία 2007 έως 2013 σε σχέση με τη Ρουμανία, 147 εκατομμύρια ευρώ ε, έχουμε διαθέσει και όπως είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση, τα χρήματα αυτά είναι διαθέσιμα και για την ενίσχυση της ε, ε, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτει και τη φυματίωση και άλλες μεταβιδόμενες ασθένειες. Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ ημών, του ECDC και του ΠΟΗ, έχουμε υπογράψει μια συνεργασία με τον ΠΟΗ της Ευρώπης, ε, είναι μια δήλωση που ονομάζεται δήλωση της Μόσχας γιατί εκεί την υπογράψαμε. Χάρτη πορείας για, πολλές στρατηγικούς, για πολλούς τομείς, για ζητήματα ε, ασφαλείας έχουμε ετησίως συνεδριάσεις με τον ΠΟΗ ε, Ευρώπη για να έχουμε για, για να ε, συνδέσουμε τις δικές μας δράσεις για τη δημόσια υγεία με αυτές του ΠΟΗ ε, και με αυτές του ECDC. Το παράδειγμα ήταν για παράδειγμα η κοινή συλλογή στατιστικών στοιχείων για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, δηλαδή ΠΟΗ, ECDC και Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή για να μην υπάρχει διπλή καταγραφή στοιχείων και να έχουμε ένα ενιαίο εργαλείο σύγκριση στατιστικών στοιχείων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Επίσης, μας ρωτήσατε για τις, τους ε, πόρους χρηματοδότησης Σε αυτό το σχέδιο δράση δεν έχουν συμπεριληφθεί ρήτρε χρηματοδότηση. Ε, βέβαια, μπορεί να υπάρχουν άλλα ε, ταμεία που μπορούν να υποστηρίξουν την προσπάθεια. Αναφέρθηκα, για παράδειγμα, σε διάφορα προγράμματα, ε, στο πλαίσιο του προγράμματο υγεία ή του ερευνητικού προγράμματο. Αν έχει κανεί ένα στρατηγικό πρόγραμμα δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί κανεί να ληφθεί υπόψη είτε υπό το πρόγραμμα υγεία ή από το πρόγραμμα έρευνα. Όσον αφορά τώρα την ε, αντίσταση ε, των, ε, στα διάφορα μικρόβια, πάλι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα αν χρειαστεί. Υπάρχει μία πρωτοβουλία με, για νέα αντιβιωτικά μαζί με την φαρμακοβιομηχανία και είναι κάτι το οποίο θα υποστηριχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας ή του προγράμματος IMI. Ε, υπάρχει ένας κατάλογος λοιπόν μέτρων που πρέπει να ληφθούν και αν χρειάζεται θα ε, ε, χρησιμοποιηθούν και τα παρέτα κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ. Ο, κύρι, ο λόγος του κύριο Σπρέγκλερ από το ECDC. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, είναι αρμοδιότητα των κρατών μερών, μερών να καταπολεμήσουν τη φυματίωση. Εγώ επισκέφτηκα πολλές χώρες όπως τη Λιθουανία και τη Ρουμανία και πραγματικά ανησυχώ πάρα πολύ. Αυτό που είναι σημαντικό στην καταπολέμηση της φυματίωσης είναι να υπάρχει ένα μηχανισμός, ένα σύστημα υγείας που να δουλεύει. Πρώτον να εντοπιστεί, στη συνέχεια να διαγνωστεί το κρούσμα. Για παράδειγμα στη Λιθουανία 20% των κρουσμάτων φυματίωσης ε, είναι πολυανθεκτική φυματίωση. Επομένως μιλάμε για ε, τεράστια ποσά για τη θεραπεία τους και δεν ξέρω εάν γνωρίζω, αν γνωρίζουν καν όλα τα κρούσματα, αν έχουν ε, εντοπιστεί τα κρούσματα και πήγα και στη Ρουμανία και εκεί το ερώτημα είναι το εξής. Έχουν αρκετά χρήματα να ε, πληρωθούν τα φάρμακα για τα παιδιά. Να σας το πω, μα, αυτό είναι το ερώτημα. Ε, είναι πραγματικά σοκαριστικό να βλέπει κανείς ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο, ότι με όλα αυτά τα μέτρα δηλαδή της λιτότητας, εγώ ελπίζω ότι οι χώρες θα μπορέσουν ακόμη να ε, έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση φάρμακα. Δεν είμαι πολιτικός, αλλά με απασχολεί πάρα πολύ. Θα ήθελα επίσης να επανέλθω στο ερώτημα της κυρίας Μέρκης, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, το κατά πόσο υπάρχει ένας ε, ε, τρόπος να ελέγξουμε την ανθεκτικότητα. Ακούσαμε ιστορίες για την, στην Ινδία ότι υπάρχει κάποιος ορισμός όχι, δεν υπάρχει ορισμός. Αν υπάρχουν έξι φάρμακα, τα δοκιμάζουμε και αν δεν δουλεύουν, τότε έχουμε μία ε, περίπτωση ανθεκτικότητας. Αν όμως έχουμε 12 φάρμακα, τότε είναι διαφορετική η κατάσταση. Οπότε κάναμε έκκληση προσπάθειας τυποποίησης αυτής της προσπάθειας, αλλά παρακαλούμε να μην ε, ε, κυκλοφορούν απλώς ε, ε, διάφορες ιστορίες. Προσπαθούμε να έχουμε μια συγκρίσιμη μεθοδολογία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην Ευρώπη και είναι γεγονό ότι είναι ανησυχητική κατάσταση. Καλό είναι να είμαστε πιο προσεκτικοί. Χαίρομαι επίση ιδιαίτερα με, αυτήν, με αυτό το blueprint για την ανάπτυξη εμβολίων. Είναι μια νέα πρωτοβουλία. Υπάρχει ένα νέο εμβόλιο κατά τη, φυμα... Υπάρχει ένα εμβόλιο κατά της φυματίωση, το οποίο δεν είναι ε, πάρα πολύ, ε, δεν δουλεύει πολύ καλά ε, υπάρχουν χρήματα για να αναπτυχθεί ένα πιο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της φυματίωσης και ελπίζουμε ότι σε πόσα χρόνια στρέφομαι προς τον δόκτωρα Μπερτολίνη, σε 5-10 χρόνια ελπίζω να το έχουμε αυτό το νέο εμβόλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε την Επιτροπή, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Επιτροπή Ελέγχου και πρόληψης ε, λιμωδών νοσημάτων. Τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, μια στιγμή να χαιρετήσω τους προσκεκλημένους μας. So, Τελευταίο θέμα της ημέρης διάταξης, προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Πρέπει να δώσουμε γνωμοδότηση στην Επιτροπή Γεωργίας. Η συγκήτριά μας είναι η συνάδελφος Λιωτάρ. Θα σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν θα πω πολλά. γιατί ήδη είναι μακριά η μέρα. Πολύ ενδιαφέρουσα σίγουρα. Θα επιχειρήσω λοιπόν να είναι πολύ σύντομη. Η γνωμοδότησή μου είναι μόνο μια σελίδα. Δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει λοιπόν πολύ. Ελπίζω να το θέλετε θετικό ότι είμαι τόσο συνοπτική. Εάν θέλετε να βελτιώσετε την προσέγγιση μου, παρακαλώ αλλά για μας το θέμα είναι να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα ως Επιτροπή Περιβάλλοντος για το όλο θέμα της μεταφοράς των ε, ζώων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση όπως είναι. Ε, και αυτό είναι το μόνο που θέλω να επιτύχω. Αν θεωρείτε ότι χρειάζονται τροπολογίες, παρακαλώ. Υποβάλλετε τροπολογίες. Υπάρχουν πολλά στραβά με τη μεταφορά των ζώων. Εξαντλούνται τα ζώα, υπερθερμαίνονται δεν έχουν επαρκή χώρο και ορισμένες φορές η ταχύτητα της μεταφοράς ε, είναι το κύριο στοιχείο και όχι η ποιότητα του περιβάλλοντος. Πολλές κριτικές λοιπόν μπορούμε να κάνουμε. Ένα από αυτό που θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη μας είναι η ανάγκη να αναθεωρήσουμε το χρόνο, τη διάρκεια των μεταφορών. Είναι το απόλυτο maximum. Ε, υπάρχει μία αναφορά με ένα εκατομμύριο υπογραφές και πάνω από τους μισούς ευρωβουλευτές έχουν ε, υπογράψει μία γραπτή δήλωση. Για το θέμα αυτό πρέπει να το συμπεριλάβουμε στην πρότασή μας. τα ζώα που μεταφέρονται προσφαγή δεν θα πρέπει να μετακινούνται για μεγάλο χρονοδιάστημα γιατί αυτό μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης χρειάζεται καλύτερη συνεργασία και επιτήρηση και επιθεώρηση όλα αυτά θα συνέβαλαν περισσότερο στην ευημερία των ζώων καλύτερες τεχνικές και επίσης πρέπει να βελτιωθούν τα ίδια τα οχήματα διότι αν υπήρχε περισσότερος χώρος και καλύτερος έλεγχος της ε, θερμοκρασίας και αυτό θα έπαιζε θετικό ρόλο. Αλλά φυσικά καλύτερο περιβάλλον δεν θα πρέπει να είναι πρόσχημα για να αιτιολογήσουν τη μεταφορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μεγαλύτερες αποστάσεις. πρέπει να δούμε πώς θα το διατυπώσουμε. Όσο συντομότερη είναι η μεταφορά, τόσο καλύτερα. Επίσης η μεταφορά σφαγίων και όχι ε, των ζών των ζώων μειώνει την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Έχουμε πολλές επιστημονικές μελέτες για το θέμα αυτό, τις οποίες τις έχει συνοψίσει η ΕΦΣΑ μεταξύ άλλων, ο Οργανισμός για την ε, Ασφάλεια και Υγιεινή των Τροφίμων. Πρέπει λοιπόν όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις μελέτες να ενταχθούν στον νέο κανονισμό στον τροποποιημένο κανονισμό. Μίλησα λοιπόν για τη σύσταση που αφορά τα άλογα. Αλλά αυτέ οι συστάσει θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και για άλλα ζώα. Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όσο με αφορά για όλα τα ζώα. Και επίση θα ήθελα η Επιτροπή, παρακαλώ, να υποβάλει μια πρόταση για να αντικαταστήσουμε τον ε, κανονισμό αυτόν. Δεν χρειάζεται να βραδιπορήσουμε με μελέτες επιπτώσεων πιστεύω ότι μπορούμε σύντομα να δράσουμε αποτελεσματικά ε, για να βελτιώσουμε αυτόν τον κανονισμό 762 και, αλλά οποιοδήποτε τροπολογίες θα ήταν ε, ευπρόσδεκτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την πάρα πολύ καλή εκθεσή της. Ε, συμφωνώ με όλα όσα μας είπε. Εγώ έχω κάποιες προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η έκθεση. Βεβαίως, χαίρομαι που διαπιστώνω ότι έχουν συμπεριληφθεί οι προτάσεις που αφορούν στον περιορισμό του χρόνου μεταφοράς των ζώων. Ε, δεν θέλω να περηφανεύομαι, αλλά εγώ ξεκίνησα αυτή την εκστρατεία που ε, συγκέντρωσε ένα εκατομμύριο υπογραφές. Προφανώς δεν το κατάφερα μόνη μου. Με βοήθησαν αρκετοί συνάδελφοι από άλλες χώρες και ε, πολλές οργανώσεις ε, φιλοζωικές. Αλλά κοιτάξτε, η το ένα εκατομμύριο υπογραφές ακόμα και με τη βοήθεια του ίντερνετ δεν είναι εύκολη δουλειά και μπορεί να γίνει μόνο εάν μπορεί κανείς να στηρίξει μια υπόθεση. Άρα δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν αλλαγή στην κατάσταση που επικρατεί. Επίσης, ευτυχώς τώρα έχουμε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, γιατί έχουμε την πλειοψηφία για τη γραπτή δήλωση επί του θέματος. Καλά λοιπόν τα πράγματα, αλλά να σας πω το εξής. Κυρία Συγήτρια, σωστά είπατε ότι δεν υπάρχουν μόνο θέματα καλής διαβίωσης των ζώων που διακυβεύονται. Υπάρχει και το θέμα της διάδοσης ασθενειών. Οι κτηνίατροι μου έχουν πει ότι αν δεν υπήρχε η μεταφορά ζών των ζώων πέρα από τα σύνορα, η διάδοση ασθενειών ανάμεσα σε ζωικούς πληθυσμούς θα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Άρα δηλαδή αυτό είναι θέμα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Επίσης, ως προς την ασφάλεια των τροφίμων, δεν ξέρω αν το αναφέρατε αυτό, κυρία εισηγήτρια, αλλά όταν μεταφέρονται τα ζώα και υποβάλλονται σε κόποση, σε στρες, αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του κρέατος. Γι' αυτό λοιπόν τίθεται και αυτό το θέμα εδώ της ασφάλειας και της ποιότητας ε, των, του κρέατος όταν ε, γίνεται ε, μεταφορά ζώων ε, έχουμε και πολλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Από το 2005 μέχρι σήμερα ο ρυθμός των χείρων που μεταφέρθηκαν συνερεκά αυξήθηκε κατά 7%. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ μια έκρηξη σε αυτές τις ε, μεταφορές, κατά 70 με συγχωρείτε της 100. Έχουμε λοιπόν πολλά ε, σωστά επιχειρήματα για να προβάλλουμε το έτοιμά μας. Και βέβαια η Κομισιόν τα τελευταία χρόνια συμπεριφέρθηκε πολύ άσχημα και ντροπή τη. Ο εκπρόσωπό τη την τελευταία φορά όταν θεσπίστηκε το νομοθέτημα είπε «Ξέρω ότι δεν είστε ευχαριστημένοι, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κατά το τέλος αυτής της, ε, της θητείας αυτής της Επιτροπής θα αποβάλουμε νέα πρόταση». Αυτό το έκανε πριν από 7 χρόνια και δεν έκανε βέβαια τίποτα, γιατί αντικαταστάθηκε από την Επίτροπο κυρία Βασιλείου. Και όταν εκείνη ήρθε ε, στην ακρόαση εδώ στο Κοινοβούλιο, τη ρώτησα «Τι θα κάνετε, θα υποβάλλετε πρόταση». «Ναι, ναι, ναι», είπε και δεν έκανε τίποτα. Δύο λοιπόν επίτροποι μας υποσχέθηκαν ότι θα καταθέσουν πρώτες και δεν το έκαναν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ντροπή. Κατά τα άλλα ε, υπάρχει αρκετή καθυστέρηση, άρα μας δόθηκε χρόνος για να προβάλλουμε την υπόθεσή μας ε, και δεν ξέρω αν πριν από 7 χρόνια θα συγκεντρώναμε την πλειοψηφία. Τώρα όμως το καταφέραμε. Γι' αυτό ας ασκήσουμε στην Επιτροπή όσο περισσότερη πίεση μπορούμε. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος και τώρα εκ μέρους των φιλελευθέρων έχει ε, το λόγο ο συνάδελφος ε, κύριος ε, Σανώνη. Ε, ευχαριστώ, ε, συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και η συγγήτρια και ο προλαλής σας. Θέλω να σας πω ότι η έκθεση της Επιτροπής ε, σχετικά με την ε, προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, ο κανονισμός αυτός έχει αρκετές ελλείψεις. Και θέλω να επισημάνω κυρίως ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε στοιχεία ελέγχου, τα οποία όμως είναι ανεπαρκή. Είναι ανεπαρκή για να προβούμε σε μία εντελεχή μελέτη του θέματος. Λείπουν κυρίως ε, στοιχεία που έχουν σχέση με τη μεταφορά των πουλερικών ε, και των ε, κουνελιών. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα κατά τη μεταφορά για την καλή διαβίωση των ζώων. Η ΕΦΣΑ λέει ότι ο κανονισμός δεν έχει ευθυγραμμιστεί με τις τελευταίες επιστημονικές, τα επιστημονικά πορίσματα όσον αφορά τη μεταφορά των αλόγων, εδώ αναφερόμαστε κυρίως στο χρόνο μεταφοράς. Όσον αφορά τώρα τη μεταφορά των πουλερικών, εκεί γίνεται λόγος για τις διαστάσεις των κλοβών και όσον αφορά τη μεταφορά των ε, κουνελιών ε, είναι ο τρόπος που μεταφέρονται αυτά. Η Κομισιόν λέει ότι δεν θέλει να τροποποιήσει τον κανονισμό, αλλά μας λέει ότι είναι απαραίτητο να έχουμε αυστηρότερη εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού. Και εδώ λοιπόν τίθεται το πρόβλημα των ελέγχων. Όσον αφορά στους ελέγχους, ε, το Γραφείο Τροφίμων και Εκτινιατρικών Θεμάτων τα τελευταία χρόνια εντόπισε πάρα πολλές ανομαλίες στα κράτη-μέλη, κυρίως όσον αφορά την καταγραφή των ταξιδίων δεν γίνονται απαραίτητοι κτηνιατρικοί έλεγχοι στα κράτη-μέλη. Η λύση λοιπόν όλων αυτών των προβλημάτων μπορεί να προκύψει μόνο εφόσον περιοριστεί ο χρόνος μεταφοράς, όπως το λέει και η συγκήτρια. Το Κοινοβούλιο στο Κοινοβούλιο υπήρχε αυτή η γραπτή δήλωση που στις 15 Μαρτίου εγκρίθηκε, άρα δηλαδή υπάρχει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο ε, και όπως είπαμε αυτή προέκυψε μετά από ένα εκατομμύριο υπογραφές ε, που τις ε, συγκέντρωσε ο άρθρος κ. Γιώργενσον από όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και ο πίνακας υπαριθμών 2 στην έκθεση που λέει ότι τα ταξίδια που απαιτούν χρόνο πάνω από 8 ώρες ανέρχονται, αντιστοιχούν μάλλον στο 32% του συνόλου των ταξιδιών. Αυτό λοιπόν το 32% του συνόλου των ταξιδιών αυτό, αν το αλλάξουμε, θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε κονδύλια. Καθότι η ίδια η έκθεση Επιτροπής, στον πίνακα υπαριθμών 5, προβλέπει και υπολογίζει ότι το κόστος προσαμογής ε, για κάθε όχημο ανέρχεται σε 11.800 ευρώ. Άρα δηλαδή αν μειωθούν αυτά τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, αυτό καταλαβαίνετε ότι θα ε, προκύψει σε εξοικονόμηση κονδυλίων. Τα στοιχεία που ανέφερα, πιο μικρά λοιπόν ταξίδια, αυτό θα διευκολύνει και τους ελέγχους. Εγώ βεβαίως ε, είμαι φυτοφάγος πρέπει να σας πω, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ε, εάν περιοριστεί η διάρκεια του ταξιδιού, θα έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τα προϊόντα που αποκτούμε από τα ζώα. Επίσης, το Γραφείο Τροφίμων και κτηνιατρικών Θεμάτων έχει μόνο πέντε ελεγκτές οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν την εφαρμογή αυτοκανισμού του στα 27 κράτη-μέλη. Καθίσατε λοιπόν σαφές ότι πρέπει να περιστεί ο χρόνος μεταφοράς και αυτό θα βοηθήσει και τους ελέγχους που θα είναι περισσότερο αποτελεσματικοί. Θεωρώ λοιπόν ότι η Επιτροπή με βάση την έκθεση και με βάση τα επιστημονικά στοιχεία οφείλει να σεβαστεί τη θέληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των πολιτών και να αλλάξει τον κανονισμό, να φέρει δηλαδή αυτόν τον περιορισμό κατά ανώτατο σε 8 ώρες στη μεταφορά των ζώων. Τώρα, σκιώδη συγγήτρια εκ μέρους του ECR, η Judy Gerling. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Τα περισσότερα υπόθηκαν ήδη και ίσως δεν σας λέω τίποτα καινούριο, αλλά θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Θερμές ευχαριστίες ε, προς την εισηγήτρια, η οποία παρουσίασε ένα ε, αντικειμενικό, μας έδωσε ένα μάθημα του πώς να παρουσιάζει κανείς μια σύντομη έκθεση. Εγώ ε, θα αντισταθώ στον πειρασμό να τροποποιήσω πάρα πολύ την έκθεση αυτή, αλλά θα ήθελα ορισμένα πράγματα να αναφερθούν, ειδικότερα για τα άλογα. Θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα πράγματα και γι' αυτό θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Πρέπει επίσης να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για την βιωσιμότητα των ζώων που ταξιδεύουν μακριά για να σφαγιαστούν. Ε, υπάρχει θέμα γεωγραφικής κατανομής των ε, ε, σφαγίων. Για παράδειγμα, ε, έβλεπα τα κινητά σφαγεία την περίπτωση των κινητών σφαγείων ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί πολλές φορές για να πάμε στα νησιά ας πούμε τα ζώα αυτά πρέπει να ταξιδέψουν δύο-τρεις ώρες εκτός από το οδικό ταξίδι που έχουν κάνει. Οπότε θα ήθελα να ε, τονιστεί αυτό το πράγμα περισσότερο. Όσον αφορά τώρα την εκστρατεία μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ντάν. Το ανέφερε, αλλά θα ήθελα για τα πρακτικά να εκφράσω και εγώ τις ευχαριστίες μας ε, σε επαφές ε, με τους συναδέλφους για να προσυπογράψουν ε, την προσπάθεια αυτή αλλά και στον κλάδο. Πολλές φορές κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από το να ακολουθούν τους, κανόνε. κανόνες. Θα θέλαμε μια παρουσίαση της δουλειάς που έχει κάνει η ΕΦΣΑ ξέρουμε ότι θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση σε αυτήν την εκστρατεία αν ορισμένοι συνάδελφοι δεν είχαν πάρει τα πράγματα τόσο κατά γράμμα. Οπότε, συγχαρητήρια Νταν, πραγματικά ήταν μια καταπληκτική εκστρατεία και αν μπορώ να κάνω οτιδήποτε για να βοηθήσω περισσότερο, ευχαρίστως. Ε, εγώ περιμένω εναγωνίως να το συζητήσουμε και να πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο, τελευταία ομιλήτρια η Πιλάρα Αγιούζο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να συγχαρώ την κυρία Λιωτάρ για την ε, τόσο σαφή και συνοπτική έκθεση που μας έκανε. Σίγουρα Αν ρωτήσουμε τους πολίτες μας αν θέλουμε να βελτιωθεί η ευημερία των ζώων, όλοι θα πούνε ότι βεβαίως να βελτιωθεί και η ευημερία των ατόμων και όλα στον κόσμο. Όσο καλύτερα είναι τα αυτοκίνητα και όσο καλύτερη είναι η θερμοκρασία και η υγρασία βεβαίως, θα βελτιωθεί η ευημερία, η κατάσταση των ζώων και των ατόμων. Όσο πιο σύντομο είναι το ταξίδι, τόσο καλύτερο είναι το ταξίδι όποιον και να ρωτήσετε αν προτιμάει να πάρει μία πτήση ε, χαμηλού κόστους ε, όπου τα πόδια του να μην χωράνε φυσικά θα σας πει ότι θέλει να είναι σε μια αντιθέση. Όλοι λοιπόν θέλουμε τα πάντα να τα βελτιώνουμε. Προφανώς. Αλλά το θέμα αυτό θα πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο του. Στην Ευρώπη έχουμε την νομοθεσία για την ευμερία των ζώων την πιο αυστηρή του πλανήτη. Από τότε που έχει εφαρμοστεί ο κανονισμός, το κόστος για τη μεταφορή θεωρούμε ότι έχει βελτιωθεί κατά 20%. Η ΕΦΣΑ λέει ότι οι συνθήκες ε, μεταφοράς είναι πιο σημαντικές από το μήκος της μεταφοράς, εκτός από την περίπτωση που αναφέρθηκε για τα άλογα. Η Κομισιόν δεν θέλει να τροποποιήσει αυτόν τον κανονισμό. Είπαμε για το διαφυγόν κέρδος που θα υπάρξει. Και ξέρετε ότι μειώνεται η ανταγωνιστικότητα της κτηνοτροφίας μας έναντι των τρίτων χωρών. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει τα ζώα να έχουν καλές συνθήκες ζωής. Αλλά αν μιλάμε για καλές συνθήκες πρέπει να κάνουμε και το διαχωρισμό μεταξύ αυτών που πάνε στο σφαγείο και αυτό που δεν πάνε στο σφαγείο πάνε για, σε ένα άλλο μέρος για να παχυνθούν κτλ. Και πρέπει να κάνουμε τις επιθεωρήσεις. Αλλά όχι μόνο για αυτά που μεταφέρουμε εντός, αλλά και για αυτά τα οποία εισάγουμε. Και αυτό έχει ως συνέπειο ότι πολλά, πολλές εκμεταλλεύσεις μετακινείται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά μας πουλάει τα προϊόντα της ακριβώς για να αποφύγει όλες αυτές τις προδιαγραφές. Πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο όλων των παραγόντων και να καταλήξουμε σε μια λύση που σίγουρα να είναι καλή για τα ζώα, αλλά καλή για την οικονομική δραστηριότητα. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην Επιτροπή να μας εξηγήσει η Κομισιόν γιατί πολλές φορές ε, δεν τήρησε τις υποσχέσεις της ε, και δεν μας υπέβαλε προτάσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ δεν έχω καλά νέα να σα ανακοινώσω, ε, γιατί γνωρίζετε ποια είναι η γραμμή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, διαβάσατε τη σχετική έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να ξαναρχίσει η συζήτηση για τον κανονισμό για την μεταφορά των ζώων. Νομίζω λοιπόν ότι όσον αφορά τις 8 ώρες ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο εδώ και πολύ καιρό ε, υπάρχει, τουλάχιστον εδώ και 12 χρόνια που εγώ δουλεύω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ακούω αυτό το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει, και υπόθηκε στην τελευταία παρέμβαση, δεν υπάρχει επιστημονική βάση για αυτές τις 8 ώρες. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η τελευταία παρέμβαση είναι πολύ πιο σωστή σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν από τους επιστήμονες, οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν είναι τόσο η διάρκεια που είναι καθοριστικός παράγοντας, όσο οι συνθήκες της μεταφοράς και πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό. Αν θέλουμε να βασιστούμε στα επιστημονικά στοιχεία, πρέπει την ευημερία των ζώων να τη βλέπουμε σαν κάτι το σφαιρικό και να μην το βλέπουμε μονοδιάστατα το θέμα. Γι' αυτό η γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο κανονισμός ε, να επιβάλλει κάποιες συνθήκες, οι οποίες βέβαια είναι πολλαπλές. Δεν είναι μόνο η διάρκεια, είναι και ο χώρος, είναι και τα οχήματα, είναι και η κατάσταση και η δυνατότητα των ζώων να μεταφερεθούν ε, γενικότερα η ευημερία των ζώων και όχι μόνο η διάρκεια. Είναι γεγονός ότι η διάρκεια έχει τη σημασία της γιατί ε, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της μεταφοράς, τόσο η μεταφορά μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα για την ευημερία των ζώων ε, όταν παρατείνεται η διαδρομή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πιστεύει ότι υπάρχει στον κανονισμό μια διαφορά μεταξύ των τεχνικών συνθήκων ε, ε μεταφοράς πέρα από μια διάρκεια 8 ε, ώρων και κάτω από τη διάρκεια των 8 ώρων, αλλά από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ε, υπόκεινται στις γενικές παραμέτρους της μεταφοράς. Ο κανονισμός επίσης αναφέρεται και στο θέμα της εκπαίδευσης των ε, οδηγών, κάτι που δεν αναφέρθηκε και είναι πολύ σημαντικό και αυτό περισσότερο από τα τεχνικά στοιχεία, γιατί η ικανότητα του οδηγού να διαχειριστεί τις συνθήκες είναι αυτή που πραγματικά δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης της μεταφοράς με καλύτερο τρόπο. Οπότε, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονεί ότι η εφαρμογή του υφισταμένου κανονισμού είναι ουσιώδης και γι' αυτό ακριβώς δίνει προτεραιότητα σε αυτές τις δράσεις. Υπάρχουν δράσεις που αναφέρονται συγκεκριμένη έκθεση. Το λέω αυτό γιατί ε, το Γραφείο Κτηνιατρικών Θεμάτων έχει 5-6 επιθερωτές. Μα δεν είναι ο ρόλο του να, να ελέγχει τη μεταφορά των ζώων αυτό το γραφείο. Ε, υπάρχει μια μικρή σύγχυση, ε, παρεξήγηση. 5-6 επιθεωρητέ ε, για να ελέγξουν ε, όλε τι μεταφορέ των ζώων στην Ευρώπη. Τι να σα πω, αυτό είναι εντελώ γελίο και ανέφικτο. Ε, πρέπει να γίνεται ένα έλεγχο των συστημάτων μέσω του γραφείου αυτού στα κράτη-μέλη. Για μένα λοιπόν το να επανδρώσουμε περισσότερο αυτό το γραφείο δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Πρέπει να δούμε κατά πόσο το κράτο μέλο έχει ένα σύστημα, ένα μηχανισμό για να ενημερώνει, ε, για να αναπτύσσει τα μέσα ε, που χρειάζονται για την ενέργεια των ελέγχων. Ο έλεγχο είναι ο ρόλο όχι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά των κρατών μελών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Εμεί είμαστε εδώ, έχουμε μια συγκεκριμένη δουλειά να κάνουμε και είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα να ε, διαθέσουν όλα τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν, όχι μόνο τις διαδικασίες επί που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τα μέτρα ενίσχυσης και πλατφόρμες συζήτησης για καλύτερη ε, κατανόηση των τεχνικών απαιτήσεων και καλύτερη γνώση και καλύτερη διάδοση των ε, καλών πρακτικών, όπως επίσης και την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για την ερμηνεία της νομοθεσίας όταν υπάρχει πρόβλημα με την κατανόησή της. Αυτό λοιπόν είναι το, ε, αυτή είναι η θεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, επίσης να επαναλάβω ότι δημοσίευσαμε προσφάτως ε, τη στρατηγική για την ευημερία των ζώων που αυτή η φιλοσοφία της ανάπτυξης ενός συστήματος ε, στήριξης, ξέρω ότι δεν είναι αντικείμενο της σημερινής συζήτησης, αλλά υπάρχει τέλος πάντων μια ευρύτερη θεώρηση ώστε όλοι όσοι ε, συμμετέχουν στη διαδικασία να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να είναι ικανότεροι να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Ε, Αν υπάρχει τώρα ένα σύστημα το οποίο μακροπρόθεσμα δεν δίνει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να δίνει, ε, τότε να το ξαναδούμε. Αλλά νομίζω ότι για την ώρα το σύστημα που έχουμε είναι πολύ πιο παραγωγικό προς τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Να δώσω άλλη μια φορά το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τις ε, παρεμβάσεις τους. Άκουσα πολύ προσεκτικά. Με χαρά θα ακούσω και τις πρωτοβουλίες και τις ε, σας. Τα συγκεκριμένα σημεία που αναφέρατε. Επίσης ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος από την Επιτροπή. Δηλαδή, ε, θα έλεγα ότι αυτά που μας είπε δεν είναι αρκετά. Γιατί επί της ουσίας ε, δεν κάνετε κάτι. Και επίσης, ε, από ό,τι κατάλαβα, θα συνεχίσετε με έναν ξεπερασμένο κανονισμό και τώρα μιλάτε για χρόνους μεταφοράς, αλλά θα πρέπει να είμαστε σαφείς. πολλοί στην Ευρώπη επιθυμούν κάποια αλλαγή και αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια δουλειά να κάνει. Πρέπει να ε, δραστηριοποιηθεί. Δεν πρόκειται για τον, ε, τη μείωση του χρόνου μεταφοράς πρόκειται για το ότι είναι ξεπερασμένος ο κανονισμός και δεν λαμβάνεται υπόψη ποια είναι τα τελευταία επιστημονικά συμπεράσματα, γιατί υπάρχουν αυτά. Υπάρχει λοιπόν ένας οργανισμός, ο ΕΦΣΑ, ο οποίος έχει δημοσιεύσει ολόκληρες εκθέσεις από αυτού του θέματος και νομίζω αυτό και μόνο αρκεί για να αποσυρθεί ο κανονισμός για να γίνει κάτι εν πάση περιπτώσει γιατί πραγματικά το βρίσκω σκάνδαλο αυτό που μας είπατε εδώ λυπάμαι πάρα πολύ, αυτή είναι η γνώμη η ο Ντάνιελ. Συμφωνώ σε μεγάλο μαθό με αυτά που είπε μόλις ο... η εισηγήτρια και να προσθέσω ότι μερικά τα προβλήματα που έχουμε με την εφαρμογή θα μπορούσαν να επιληθούν αν απλοποιούσαμε κάπως την νομοθεσία. Ένας από τους λόγους που είναι τόσο δύσκολο να ελέγξουμε και οι μεταφορείς να εφαρμόσουν τον κανονισμό είναι ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι κανόνες, πώ να πάρει ε, το ζώο, να το βάλει στο αυτοκίνητο, πώ πρέπει να περιμένουν, πότε πρέπει να το ξαναβάλει στο αυτοκίνητο, στο φορτηγό. Εάν μειώσουμε το χρόνο μεταφορά, θα είναι πολύ πιο εύκολο να ε, ελέγξουμε και να εφαρμόσουμε. Αλλά τώρα δεν θα μπω τώρα σε όλα τα τεχνικά επιχειρήματα που ανέφερε η Κομισιόν, αν και έχω αντεπιχειρήματα. για σχεδόν όλα. Να ακούω τώρα την Κομισιόν να λέει ότι δεν υπάρχει επιστημονική επιχειρηματολογία για να μειωθεί ο χρόνος μεταφοράς. Απίστευτα. Οποιοςδήποτε επαγγελματικά ασχολείται με αυτό μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι έτσι έχουν τα θέματα. Εν πάση να κάνω μια ερώτηση. Δύο επίτροποι δήλωσαν και θα μπορούσα να βρω και τα πρακτικά τα έχω και σε βίντεο ίσως. Δύο επίτροποι είπαν ότι ήθελαν αναθεώρηση της νομοθεσίας. Ερώτηση λοιπόν. Τι έχει αλλάξει. Και τώρα ξαφνικά δεν θεωρείται ότι χρειάζεται αναθεώρηση. Ευχαριστώ κύριε Γιώργενσεν. Έκλεισε η συζήτηση. Πρέπει να πω Ενδιαφέρουσα παρουσίαση ε, είδαμε εδώ από την Κομισιόν. Μέχρι στιγμής δεν έχω ασχοληθεί σοβαρά με την ε, προστασία των ζών. Μπορώ όμως ότι μετά από αυτή την παρουσίαση σας σήμερα θα ασχοληθώ. Και ότι εκείνοι οι οποίοι συγκέντρωσαν ένα εκατομμύριο υπογραφών γελάτε. Δεν ξέρω γιατί το θεωρείτε τόσο αστείο. Πρέπει να σας πω ότι όλοι όσοι συνέλεξαν ένα εκατομμύριο υπογραφών θα ήθελα να τους ε, προσκαλέσω από 1η Απριλίου 2012 να αναλάβουν μια πρωτοβουλία πολιτών και να χρειαστεί να δολογεδίσετε. Ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω. Πρέπει να το πω. Και επειδή έγινε μια ερώτηση, ε, παρακαλώ απαντήστε. Όσο αφορά τις δεσμεύσεις των προηγουμένων επιτρόπων, δεν έχω συγκεκριμένη ε, ανάμνηση, αλλά κα, καμιά φορά υπάρχει κάποια σύγχυνση. Ο Επίτροπος έχει το χαρτοφυλάκιό του, αλλά οι αποφάσεις που λαμβάνονται, λαμβάνονται από το σώμα των Επιτρόπων. Μπορεί να υπάρξουν διαπραγματεύσεις κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ένας Επίτροπος μπορεί να έχει τη βούληση να θέλει να κάνει κάτι, αλλά στα πλαίσια της Κομισιόν μετά μπορεί να γίνουν εσωτερικές συζητήσεις Πρέπει να καταλάβετε ότι λαμβάνουμε υπόψη την ε, επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, αλλά υπάρχουν και άλλες απόψεις που λαμβάνονται υπόψη όταν λαμβάνει απόφαση η Κομισιόν. Ένας ευρωβουλευτής, μία ευρωβουλευτής, μίλησε για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και μπορεί μετά η διαπραγμάτευση να δώσει διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν έκανε τίποτα για τα 7 χρόνια. Δεν είναι αλήθεια. Υπήρξε μία εργασία εξέταση του θέματος. Αυτό Μπορεί να μην έχει νομοθετικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγινε τίποτα. Έγιναν ορισμένα πράγματα, αλλά τα οποία δεν οδηγούν σε αναθεώρηση της νομοθεσίας. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ε, έχω κίνητρο για να ασχοληθώ με το θέμα αυτό και θα τα ξαναπούμε κατάλληλη, στο κατάλληλο πλαίσιο για το θέμα αυτό. Διακόπτεται η συνεδρίαση. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10 για τη συνέχιση των εργασιών μας. Ευχαριστώ. Α,